myself. Thank you. I think we'll start the meeting. Καλησπέρα σε αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως και εγώ και μερικοί άλλοι κολλήσαμε σε διάφορα σημεία λόγω του χιόνιου και της κακοκαιρίας. Εν πάση περιπτώσει, αρχίσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ο εισηγητής και πολλοί σκιώδη εισηγητές ζήτησαν αναβολή της ψηφοφορίας για τη ε, σχέδια έκθεσης για το CCCBTB. Συμφώνησα με την αναβολή της ψηφοφορίας για τις 20 και 21 Μαρτίου στην συνεδρία του Μαρτίου. Έχω μερικές ανακοινώσεις. Καταρχήν, οι αιτιολογημένες γραμματοποίησεις ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων για τη μη συμμόρφωση με το σχέδιο νομοθετικής πράξης ως προς την αρχή της επικουρικότητας έχουν κοινοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στο, στην προθεσμία των 8 εβδομάδων του άρθρου 8 παράγραφος 2 της Συνθήκης Λισαβόνας για το θέμα αυτό και έχουν δημοσιευθεί στο σημείο 4 της ιστοσελίδας στα πλαίσια του σημείου 4 της ημερήσια διάταξη. Κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τι δραστηριότητε των εταιριών. Έχουμε και τη διόρθωση για τη νομοθεσία για το short selling. Νομοθετική, νομική μάλλον διόρθωση. Οπότε τον νέο αναθεωρημένο κείμενο μετά τη γλώσσα, την γνωμάτευση νομικής υπηρεσίας θα δημοσιευθεί με βάση το ε, κανόνα 2161 του των διαδικαστικών κανόνων και στην μερική ε, ολομέλεια του Φεβρουαρίου θα θεωρηθεί ως συγκεκριμένη εκτός και αν κάποια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 βουλευτές ζητήσουν να γίνει ψηφοφορία επί του διορθωτικού παρόλο που είναι μόνο νομική διόρθωση. Σε ό,τι αφορά το τριμερή διάλογο για τα, για τα παράγωγα, ο έκτος τριμερής διάλογος έγινε στις 30 Ιανουαρίου, σημειώθηκε κάποια πρόοδος και απέμεινε εκρεμές ένα μόνο ουσιαστικό πολιτικό ζήτημα. Και τελευταίος τριμερής διάλογος θα γίνει στα τέλη της εβδομάδας, ίσως πέμπτη αργά το απόγευμα. Περιμένουμε ακόμη την επιβεβαίωση της ε, ημερομηνίας. Αυτά ως προς ανακοινώσεις. Περνάμε στο σημείο 3, διαχείριση ποιότητας στον τομέα των ευρωπαϊκών στατιστικών. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Έντβαρτ Σικλούνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε ε, παρά να αναγνωρίσουμε τη μεγάλη σημασία της ε, διαχείρισης ποιότητας των μέτρων ευρωπαϊκών στατιστικών να δούμε τι γίνεται με το Six ε, τη συνθήκη, την Ατζένα 2020 και το λεγόμενο scoreboard. Ε, βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι αν δεν είναι ισχυρή η βάση και μπορεί να υποστηρίξει όλα τα συμπεράσματα, όπως ξέρουμε. Θα βρισκόμαστε πάνω σε ανασφαλές έδαφος και θα έχουμε προβλήματα. Αυτή η έκθεση λοιπόν έχει σαν στόχο να τονίσει τη σημασία της ενδυνάμωσης εκείνων των ε, οργανισμών που προετοιμάζουν τα στοιχεία. Ιδίως όσον αφορά την εξαρτησία τους. Είναι σημαντικό οι κυβερνήσεις να μην άπτονται αυτών των οργανισμών Και αυτοί οι οργανισμοί, όπως και μια κεντρική τράπεζα, θα πρέπει να τη χάνουν σεβασμού και να κερδίσουν την αξιοπιστία τους εφόσον είναι πραγματικά ανεξάρτητες. Να ασκούν ισχυρή διακυβέρνηση κατά την ε, συλλογή, προετοιμασία, ταξινόμηση και δημοσία των στοιχείων, να ακολουθούν κάποιο κώδικα συμπεριφοράς και οι εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι που χρειάζονται λαμβάνουν χώρα. Γίνεται διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών. Και το Ελεκτρικό Συνέδριο ζητά έντονη δέσμευση και από τις κυβερνήσεις που χρηματοδοτούν και από, τις ίδιες, από τους Αντεστώντα τα στοιχεία αυτά, βλέπουμε ότι η κύρια πηγή είναι οι κυβερνήσει. Με τα στοιχεία για τα δημόσια οικονομικά. Και εδώ θεωρούμε τις κυβερνήσεις υπεύθυνε να δίνουν βάσιμα στοιχεία κάτω τη δυνατόν και τυποποιημένα και συγκρίσιμα στοιχεία έγκαιρα. Ξέρουμε ότι στο παρελθόν αυτό ήταν πηγή προβλημάτων στην Ευρωζώνη. Και αυτό είναι ένα σημείο που τονίζει ιδιαίτερα. Όσον αφορά μικρές χώρες, ε, όχι μικρές δηλαδή, ιδίως αδύναμες θα ήθελα να πω, όπου υπάρχουν ε, ε, εξαιρέσεις και αποκλήσεις όσον αφορά την χορήγηση των στοιχείων. Αυτό μπορεί να είναι καλό αφενός, αλλά αφετέρου σημαίνει ότι λείπουν κάποια από τα στοιχεία και οι χρήστες υποφέρουν από αυτό. Γι' αυτό δεν περιμένουμε η Κομισιόν να δώσει χρήματα, αλλά το στράσιο να προωθεί τις απαραίτητες ε, τεχνογνωσίες, ώστε να υπάρχουν ισχυρά στατιστικά στοιχεία. Όσον αφορά τη δημοσίευση, λέμε ότι θα πρέπει να είναι φιλικά προς το χρήστη τα στοιχεία αυτά ακόμα και για άτομα χωρίς τεχνικές γνώσεις και επίσης για τους πολιτικούς. Όπως ξέρετε, και οι κυβερνήσεις και άλλοι θέλουν μόνο τους να ερμηνεύουν τα στοιχεία αυτά και θα πρέπει να φτάσουμε σε στη στο οποίο ο χρήστης, οποιοδήποτε να είναι και αυτός, να μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά άμεσα και όχι να τα παίρνει από άλλες δευτερεύουσες πηγές. Να μην χρειάζεται δηλαδή ε, κάποιος ε, ιδιαίτερα ειδικευμένο για την επεξεργασία των στοιχείων αυτών που υπάρχουν online. Και τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να χορηγούνται χώρα προς χώρα όπου είναι δυνατόν. Και είναι μια γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης η οποία θα έλεγα είναι απόλυτα αποδεκτή. Σε γενικές γραμμές λοιπόν οι ομάδες από κοινού συγχώνησαν πάνω σε μια σειρά συμβαστικών τροπολογιών που ελπίζω θα τύχουν τις πλήρες υποστήριξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θα ήθελε να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Ο που σιάζει σε αφουσιάζει Σβέν. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον υπάρχουν άλλε ομάδε που θέλουν να μιλήσουν πριν από μένα. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σιγκλούνη για την πολύ καλή συνεργασία και να τονίσω ότι στην έκθεση και στο συμβιβασμό θα μπορέσουμε να τονίσουμε, όπως είπατε και εσείς, να αυξήσουμε την ε, ε, εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία αυτά της Ευρωστάτ. Όπως είπατε και εσείς, έχει βελτιωθεί η Ευρωστάτ από σχετικά με το παρελθόν. Και τώρα γίνεται άλλο ένα βήμα προς τα εμπρός. Δηλαδή θα πρέπει τα στοιχεία αυτά να είναι διαθέσιμα ούτως ώστε όλες οι χώρες και όλοι οι πολίτες των χωρών να έχουν εντύπωση ότι έχουν πρόσβαση αυτά τα στοιχεία. Και επίσης είναι καλό να υπάρχουν γραφικές παραστάσεις στην ιστοσελίδα της Eurostat, όπως το κάνουν και άλλοι σχετικοί οργανισμοί. Η Ευρωστάτη έδωσε το καλό παράδειγμα όταν ε, δημοσίευσε τα στοιχεία για το χρέος, ακόμα και είχε αμφιβολίες για το βάσιμο των στοιχείων αυτών των εθνικών οργανισμών. Ε, συμφωνούμε νομίζω με τον εισηγητή ότι θα πρέπει η Ευρωστάτη να το κάνει αυτό πιο συχνά, ούτως ώστε να είναι απόλυτα διαφανές και ανοιχτό κατά πόσον τα στοιχεία που υπάρχουν δείχνουν να είναι βάσιμα ή όχι, κατά πόσον υπάρχουν αμφιβολίες, κατά πόσον υπάρχει ανάγκη βελτίωσης του τρόπου με τον οποίο προετοιμάζονται τα στοιχεία αυτά από τους εθνικούς οργανισμούς. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ και θα ήθελα στον λόγο για την διαχείριση ποιότητας των ευρωπαϊκών Α, ναι, ωραία. Θα ήθελα να απαντήσω στα σχόλια του Σφέν. Δεν θα υποστηρίζω την τροπολογία του 25 και 26, γιατί εμείς έχουμε υποβάλει τροπολογία 27 και 28. Δεν είναι ότι οι παρατηρήσεις του δεν είναι σωστές αλλά είναι πολύ παρόμοιες με τις που κάνω εγώ στη δική μου τροπολογία παρελθόν 35 για την καλή ισορροπία μεταξύ του επίκαιρου της ποιότητας των πληροφοριών. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σίγουροι ότι όταν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες, οι πληροφορίες αυτές να είναι υψηλής ποιότητας και ακρίβειας. Και όχι μόνο επίκαιρες. Καμιά φορά δεν μπορούν να συλληφθούν τα στοιχεία τόσο γλυγρό όσο θα ήθελε κανένα. Αυτό λοιπόν είναι μία παρατήρηση. Και είπατε υποστηρίζω την δική σας τροπολογία όσον αφορά την ε, αποκάλυψη της ε, ε, ευθύνης των, της των στοιχείων. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή και όταν εξετάσουμε τη δική σας έκθεση Σάρα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να εντάξουμε τα στοιχεία αυτά επίσης. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή ε, γιατί συμμερίστηκε αν θέλετε το βάρος των στατιστικών που αυτή τη στιγμή ε, είναι μοιρασμένο σε πολλούς ε, εισηγητές εδώ στο Προεδρείο. Σοπόλης, τυπικά σκιώδης εδώ. Θες το λόγο, όχι. Άλλος. Όχι, δεν έχω ερωτήσει, δεν έχω σχόλια. Όλα, όλα καλά. Ωραία, η έκθεση είναι καλή. Πολύ ωραία. Θαυμάτια. Θα ψηφίσουμε σύντομα. Α, συγγνώμη κύριε Χούντι, δεν σας είδα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που χαλάω λίγο τη ροή, αλλά είχα ζητήσει το λόγο. Βεβαίως σε λίγο θα ψηφίσουμε και επομένως ε, ε, κρίνοντας και με βάση τη voting list, επιτρέψτε μου γιατί έχει τη σημασία να επιμείνω σε δύο-τρία σημεία. Έχουμε καταθέσει σχετικές τροπολογίες. Ε, βλέπω ότι ο εισηγητής δεν τις εστερνίζεται. Επιτρέψτε μου λοιπόν δύο παρατηρίου, τρεις παρατηρήσεις. Το, η πρώτη παρατήρηση έχει σχέση με την τροπολογία για κάποιον που είναι σχολαστικός 6. Στο σημείο όπου η εισήγηση ισχυρίζεται δικαίως βεβαίως ότι η κρίση δημιουργεί τον πειρασμό να δημιουργηθούν απάτες και αλχημίες στη στατιστική. Κατά τη γνώμη μου, όπως είχα πει και την άλλη φορά και θα σας δώσω και κάποια στοιχεία, εδώ υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα. Και πριν την περίοδο της κρίσης, η επεξεργασία και η ανοχή των στοιχείων και εκ μέρους της Eurostat, όχι των μεμενωμένων χωρών, αποδεικνύονταν ότι είχε λαθροχειρίες ή ανοχές. Θυμίζω την ακρόαση που είχαμε κάνει για τα περίφημα swaps στην Ελλά... για τις... της Ελλάδας, νομίζω ήταν το Μάρτιο του 2010 κυρία Πρόεδρε, όπου αποδείχθηκε ότι αυτή την πρακτική την ακολουθούσαν και άλλες χώρες. Ήταν μια γενικευμένη νόμιμη μεν, αλλά όχι ηθική κατά τη διατύπωση που έκανε και ο Επίτροπος τότε στην περίπτωση αυτή. Η Eurostat δεν έδωσε εξηγήσει γιατί το ανεχόταν ή και γιατί το κάλυπτε. Επομένως υπάρχει θέμα ευθύνης και πολιτικών σκοπιμοτήτων όχι μόνο στην περίοδο της κρίσης που σωστά λέει η εισήγηση ανεβαίνουν οι πειρασμοί, αυξάνονται οι πειρασμοί να αλλοιώσει τα στατιστικά στοιχεία. Το δεύτερο είναι η πρόταση συμπλήρωση, δεν είναι βέβαια το κύριο θέμα του ζητήματος, ότι στους δείκτες καλό είναι να τονίσουμε ότι πρέπει να παρακολουθούνται και οι δείκτες οι οικονομικοί και περιβαλλοντικοί. Έχουμε κάνει μια γενικότερη συζήτηση σχετικά με το ΑΕΠ και άλλους τέτοιους οικονομικούς δείκτες, δεν νομίζω ότι θα δυσκόλευε αν δεχόμαστε αυτή την προσθήκη και αναφέρομαι σε αυτή την τροπολογία. Και το τελευταίο. Αυτό συμφωνώ και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε για την ανεξαρτησία των αρχών που επεξεργάζονται τα στατιστικά στοιχεία. Όμως το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται αυτή η προσπάθεια ανοίγει πόρτες για πολιτικές παρεμβάσεις. Τελειώνω λέγοντας ότι το θέμα των στατιστικών στοιχείων βρίσκεται στο επίκεντρο της Ελλάδας τώρα οι οικονομικοί ελεκτές έχουν καταθέσει πόρισμα στη Βουλή ότι αλλοιώθηκε το έλλειμμα του 2009 φούσκωσε από πολιτικά πρόσωπα και παραπέμπουν ή ζητούν να τεθεί το θέμα όσο αφορά την πολιτική ευθύνη. Εκεί έχει βάλει το χεράκι της και η Eurostat και δεν ξέρω τι προβλέπεται ή πώς θα μπορούσε να γίνει ε, στη συνέχεια ε, νομίζω ότι μια ακρόαση, αν είναι κάποιο εκπρόσωπο τη Eurostat κάποια στιγμή σχετικά με τον τρόπο που δουλεύει, με τον τρόπο που παρεμβαίνει, για να εξασφαλίσουμε αυτά που λέει η εισήγηση και ο, ο εισηγητή, την ανεξαρτησία και να μην έχουμε πολιτικέ παρεμβάσει, θα ήταν βοηθητικό. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, Εγώ Θα ήθελα να απαντήσω στον Έλληνα συνάδελφο επί τον ετών καταβλήσαν προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συλλεχθούν στοιχεία από τα κράτη-μέλη. Και αυτό παρεμποντήθηκε. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είπανε εμείς δεν επιτρέπουν τι Βρυξέλλες να μας δώσουν ενδεικτικό. Ή όπως είπε ο καγκελάριος τότε δεν θέλω να με βάλει τιμωρία οι Βρυξέλλες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στατιστικών Στοιχείων ήταν ένας οργανισμός ε, έτσι παραδιπλανός θα έλεγα, χωρί τι αρμοδιότητε που έπρεπε να έχει. Και η κρίση το κατέδειξε αυτό ξεκάθαρα. Αν θέλουμε να συνεργαστούμε χρειαζόμαστε στοιχεία βάσιμα. Χρειαζόμαστε μια ανεξαρτησία που να επιτρέπει τα στατιστικά στοιχεία να μπορούν να ελέγχονται. Αυτό μπορεί τώρα να εγγυηθεί η Ευρωστάτ, αν μπορεί να παρέμβει, να συγκρίνει και να δώσει και συστάσεις. Αυτή είναι η βασική ιδέα που θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Εάν θέλουμε να παίξουμε από κοινού, πρέπει να έχουμε κοινού κανόνε οι οποίοι να τυχάνουν χάνουν κάποια εποπτεία. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη δυνατότητα συλλογή των στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει αυτών μπορούμε νομίζω να προσπαθήσουμε να δράσουμε. Και αν το τηρήσει η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Αλλά ας τηρήσουν όλοι τους κοινούς αυτούς τους κανόνες και ας φροντίσουμε όλοι η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία να έχει τα στοιχεία αυτά στα χέρια της, στοιχεία που ξέρουμε ότι είναι σύμφωνα με την πραγματικότητα και όχι ότι απέχουν από την πραγματικότητα. Δεν θέλουμε τα κράση μέλη να μας δώσουν στοιχεία έτσι μόνο για να κάνουν ε, εντύπωση αλλά πραγματικά στοιχεία. Και αν ακολουθήσουμε αυτή την άκουσα θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη Ευρώπη. Όλα τα άλλα θα ήταν εσφαλμένα. Κύριε Σιγητά, νομίζω ότι μας δώσετε μια καλή βάση πάνω στην οποία μπορούμε να εργαστούμε. Και αυτό μπορούμε νομίζω να το διαδώσουμε και στους πολίτες των χωρών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε σε ένα λεπτό πραγματικά επί του σημείου αυτού και θα πάει στην Ολομέλεια στην πρώτη ολομέλεια του Μαρτίου πιο συγκεκριμένα. Έντουαρντ, μπορείς να ξαναπάρεις το λόγο. Μία σύντομη απάντηση στον κύριο Χουντή. Από τις τρεις τροπολογίες συμφωνώ με μία. Και είναι κρίμα που δεν συναντηθήκαμε πριν για να συζητήσουμε και τι υπόλοιπε δύο. Γιατί είμαι σίγουρο ότι με κάποιε αλλαγέ στη διατύπωση θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνήσει. Πάντω εγώ θεωρούσα... Συμφωνώ με τι ε, περιβαλλοντικέ στατιστικέ. αλλά όμω η διατύπωση που χρησιμοποιείται είναι λίγο αμφίσιμη. Γιατί η Eurostat δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση να υπερασπιστώ κάποιο θεσμικό όργανο, αλλά από ό,τι ξέρω όταν είχαν την εντολή. Ούτε από το Συμβούλιο για να ελέγξουν τα στοιχεία των δημοσίων λογαριασμών, τα δημόσια οικονομικά. Και ξέρω ότι δεν είχε πρόβλημα μόνο μία χώρα με αυτά τα στοιχεία, αλλά πολύ περισσότερες είχαν ανακριβή στοιχεία. Πολύ ωραία. Τώρα περνάμε στην ψηφοφορία. Και όπως είπα στην αρχή, για το CCTB, για το ΚΕΒ και η ψηφοφορία αυτή αναβάλλεται. Έτσι λοιπόν θα έχουμε κάποιο χρόνο στη διάθεσή μας για την κοινή δηλαδή ενωπημένη φορολογική βάση δραστηριότητα των εταιριών. Για την διαχείριση της ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών, α, δύσκολο θέμα, ε, μπορούμε να τα καταφέρουμε και χωρίς την κάρτα σου, Πασκάλ. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε τέτοια δύσκολη θέση όμως. Ίσως κερδίσουμε μάλιστα λίγο χρόνο, επειδή εκ θα ψηφίσουμε το πρώτο σημείο. Επομένως, αμέσως μετά την ψηφοφορία αυτή θα πάμε στην ε, έκθεση για την κατάχρηση της αγοράς. Αμέσως μετά την ψηφοφορία. Το λέω για όσους δεν το ξέρανε. Σον Πολ, είσαι έτοιμος για το σημείο 5. Ζητώ συγγνώμη που ζητώ το, το λόγο γι' αυτό. Μας λέτε εσείς οι υπηρεσίες σας, οι τεχνικές υπηρεσίες, τι να γίνει με το, με το κουτί μου αυτό, το κουτί του ήχου που δεν λειτουργεί καλά. Ε, είναι όπως οι αλοκαθαριστήρες στο Βέλγιο που δεν δουλεύουν καλά. Πέστε, εσείς ή πέστε τέλο πάνω στις υπηρεσίες σας, τεχνικές υπηρεσίες που ασχολούνται με τον ήχο, ότι υπάρχει πρόβλημα. Το μηχάνημά μου χάλασε. Χρειαζόμαστε ένα τεχνικό. Να βοηθήσει τον Ζαν γιατί θέλει να ακούει τη διερμηνία για να μπορέσει να ψηφίσει. Εντάξει, καταλα... ακούτε τώρα. Όταν ψηφίζουμε δεν έχω πρόβλημα, γιατί τα αγγλικά μου φτάνουν μέχρι να καταλάβω τα δικά σας όταν ψηφίζουμε. Θα δούμε, εν πάση περιπτώσει, αν το μηχάνημά σας λειτουργεί. Όλο το σύστημα του ήχου, αν λειτουργεί. I say something, are you getting Μιλάω τώρα, με ακούτε από τη διερμηνία. Ακούτε τη διερμηνία σας. Ε, κάτι πιο σοβαρό είναι. Κάποιος σαμποτάζ, κάποιος σαμπόταρε. Σαν Ναι, ναι, ναι, σαμποτάζ είναι. Δεν είναι απλό πρόβλημα με τον ήχο. Τι Καλά, εντάξει, να μου σαμποτάρει το μικρόφωνο δεν πειράζει, αλλά όχι και να με προσβάλλετε και να με βρίζετε. Okay, do we want to test that for whether we have any interpretation? Να τσεκάρουμε τη διερμηνία. Ανακούγεται. Βλέπουμε ένα τεχνικό, ο οποίο παίζει με τα μικρόφωνα εκεί και με το σύστημα ήχου. Εμεί θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ενώ οι τεχνικοί προσπαθούν να λύσουν το τεχνικό πρόβλημα του ήχου. Ζωάν Πολ, και άλλο πρόβλημα έχεις. Θέλω να μου επιτρέψετε να ψηφίσω χωρίς κάρτα, γιατί την ξέχασα. Ό, αν χρειαστεί να ψηφίσουμε με κάρτα θα μας απασχολήσει αυτό το θέμα. Προς το παρόν αφήστε το. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Περνάει. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Περνάει. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 με προφορική τροπολογία από τον εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Θα ασχοληθούμε με τη 15. Τροπολογία 15. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 1 για την τροπολογία 16. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αντί για την 16, έτσι. Η 17 καταπίπτει. Όχι. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. συμβιβασμός α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και μετά περνάμε στην 20. Όχι, λάθος. Στην προφορική τροπολογία 2 πάμε, που καλύπτει την 20. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αρχικό κείμενο παράγραφος 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός Γ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γνωμοδότηση Ρέτζι 1-5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αναφορές 1-3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, εκτιμώντας γ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβασμός δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 5 κατά αποχές εγκρίνεται,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 Τροπολογία 11 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το κείμενο πώς τροποποιήθηκε. Δεν χρειάζεται να μετρήσουμε γιατί έχουμε αρκετούς χωρίς κάρτες. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Τέλο πάντων, θα μετρήσουμε μετά του ανθρώπου χωρί κάρτα. Κλείνει η ψηφοφορία. 29 υπέρ, δύο εποχές. Πόσοι είναι χωρίς κάρτες? Πέντε. Πέντε. 34 υπέρ και δύο εποχές. Συγχαρητήρια στον συγητή. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε την ψηφοφορία. Σύντομη. Γιατί αναβάλαμε το προηγούμενο θέμα. Όσοι θέλετε να φύγετε, σας παρακαλώ γρήγορα και ήσυχα. Για να πάμε στο σημείο 6 και 7. Για την κατάχρηση της αγοράς. Η χειραγώγηση της αγοράς. Ευχαριστώ. Ησυχάστε παρακαλώ για να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. να ηρεμήστε. Για να μην υπάρχει αμφιβολία. Έχουμε και τις κάμερες εδώ. Το ζητήσαμε και εγκρίθηκε. Αρλίν. Ευχαριστώ, Σάρον. Είναι η πρώτη συζήτηση, αγαπητοί συνάδελφοι, να ανακεφαλαιώσω τι προσπαθεί να πετύχει ο κανονισμός και η οδηγία. Είναι μια αναθεώρηση της οδηγίας του 2003 MAD, να την κάνει από οδηγία κανονισμό και να εφαρμόστε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση Υπάρχει και μια νέα οδηγία που θα μιλάει για ποινικέ κυρώσει, για σοβαρέ ε, παραβάσει ε, χειραγώγηση αγορά. Και θα πρέπει οι χώρε οι οποίε δεν έχουν ποινικέ κυρώσει να ανέβουν, να ανεβάσουν την πάρα και να αποκτήσουν. Είναι βασικό τμήμα τη ε, μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να υπάρχει εμπιστοσύνη στι αγορέ. Και όπω είδαμε, και από τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο των χρηματαγορών ε, τώρα ε, με τις νέες δυνατότητε, οι δυνατότητες χειραγώγης αγοράς έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Όλα αυτά τα κενά λοιπόν, με αυτή την μεταρρύθμιση θέλουμε να τα καλύψει. Ε, όλα αυτά τα κενά που υπήρχε ε, υπήρχαν στην οδηγία MAD και στην οδηγία για, τα, για τον εξοχρηματιστριακό κύκλο και δραστηριότητες, θα τα καλύψουμε. Θέλουμε οι ρυθμιστικέ αρχέ να καταπολεμήσουν τη χειραγώγηση αγορά και η ανασφάλεια δικαίου θέλουμε επίση να πάψει να υπάρχει, να υπάρχουν δηλαδή τώρα και ποινικέ και διοικητικέ κυρώσει. Υπήρχαν μόνο ε, διοικητικέ μέχρι τώρα. Και θέλουμε να μειώσουμε το βάρο ε, για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Μια απόπειρα δηλαδή τουλάχιστον. Οι βασικέ αλλαγέ στην τρέχουσα νομοθεσία αφορούν το πεδίο εφαρμογή, ε, του ορισμού οι ορισμοί είναι ένα θέμα που προκύπτει στις συζητήσεις με τους ενδιαφερομένους. Μέτρα για να βελτιώσουμε την πρόληψη και ανείχνευση της χρειακής αγοράς και να υπάρχει, να παρεμποδίζουμε τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες οι αρχώδιες αρχές και, όπως είπα, ποινικέ και διοικητικές κυρώσεις μέσα σε αυτές τις αρμοδιότητες. Τώρα πολύ σύντομα. Θέλω να σταθώ σε κάποια από τα θέματα που θέσαμε στο γύρο τραπέζης που είχαμε με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ρυθμιστικές αρχές και τι προέκυψε από την ακρόαση. Θα συνεχίσουμε το διάλογο και με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και με τους ενδιαφερομένους για να αυξήσουμε την κατανόηση που έχουμε για αυτά τα θέματα, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει και φυσικά προσπαθούμε να χωνέψουμε αυτές τις πληροφορίες που προέκυψαν, που μας δώσανε. Και πριν περάσω στην ε, σύνταξη του κειμένου, θα την κάνω ευθέτω το χρόνο, πρέπει να τα χωνέψω αυτά. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, είναι σαφέ ότι πρέπει να καλύψουμε τα χρηματοπιστωτικά μέτρα στον εξοχρηματιστριακό κύκλο βέβαια και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 2 ε, για τις σημαντικές πληροφορίες, ο ορισμός των σημαντικών πληροφοριών. Αυτό το σημείο προέκυψε ε, σε πολλά από τα σχόλια και από τον κλάδο και από τους ενδιαφερομένους, γιατί ένας ορισμός άλλαξε και δεν καλύψει συγκεκριμένες πληροφορίες, όλες τις πληροφορίες, αλλά σημαντικές πληροφορίες. Ορισμένοι λένε, ορισμένοι, ορισμένοι εκπρόσωποι του κλάδου να λένε ότι πρέπει να διαγράψουμε αυτόν τον ορισμό που είναι πολύ ευρύς. Αλλά στην αρχική συζήτηση που είχα, ε, είπα ότι πρέπει να βρούμε μία ισορροπία, ούτω ώστε οι ρυθμιστικέ αρχέ να καταπολεμούν πραγματικά την χειραγώγηση τη αγορά και να δούμε τελικά τι είναι οι σημαντικέ ε, εμπιστευτικέ πληροφορίε, γιατί χρειάζονται αυτέ οι παραπάνω πληροφορίε για τι ρυθμιστικέ αρχέ, ούτω ώστε να καταπολεμούν την χειραγώγηση. Επίση, ε, κάποιοι μίλησαν για την έλλειψη διατάξεων για να εξασφαλίσουν την διασυνοριακή εποπτεία. Είναι ένα θέμα και στι συζητήσει που είχαμε με τι ρυθμιστικέ αρχέ προκύπτει ότι τα διασυνοριακά προβλήματα αυξάνονται. Ε, Μερικέ φορέ η πληροφορία την ψάχνουμε σε 7 διαφορετικά κράτη-μέλη, μα είπε κάποιο. Το θέμα είναι πώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και οι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ ε, θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη διασυνοριακή δραστηριότητα είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και θέλω να ακούσω τις απόψεις των σκιωδών ε, εισηγητών εδώ πριν πάρω οριστική απόφαση. Ε, τώρα, για τα OTF, ε, τους οργανωμένους μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, πρέπει να μπορούμε να εντοπίζουμε και εκεί τις ε, καταχρήσεις. Είχαμε την οδηγία MIFID, ε, μπορεί να αποφασίσουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο μηχανισμό οργανωμένης διαπραγμάτευσης, ε, αλλά αυτό θα δυσκολέψει περισσότερο τις ρυθμιστικές αρχές και θα κατακαιρματιστεί περισσότερο η αγορά. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρχει συνέπεια με τις προτάσεις MIFID, τις οδηγίες MIFID. τη οδηγία για τις αγορέ χρηματοπιστωτικών μέσων. Δεν ζητήσαμε μια νέα κατηγορία οργανωμένη διαπραγματεύση. Πρέπει να έχουμε ένα πραγματικό καθεστώς για να καταπολεμήσουμε την χειραγώγηση αγορά σαν πιο κατακαιρματισμένε οι δομέ. Επίση, ε, για το εμπόριο υψηλή συχνότητα. Μπορεί να δυσκολεύσει περισσότερο την ανείχνευση της ε, χειραγώγησης αγορά και θα πρέπει να δούμε και την έκθεση IOSCO που μιλάει για κάποιου τομεί που όπου εκείνο είναι αποτελεσματικό. Θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματικότητα τη αγοράς, ακεραιότητα και αντοχή των αγορών. Αυτά τα τρία σημεία λέει. Θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Δεν θέλουμε μέσω αυτού να μπουν νέε πρακτικές χειραγώγηση τη αγοράς. Θα πρέπει ε, αν μεγαλώσει ε, η δραστηριότητα των, του κλάδου των ενδιαφερομένων, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ανοιχνεύσουμε το πρόβλημα. Όσο υπάρχουν επίσης τεχνολογικές ε, εξελίξεις, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το high frequency trade, με το εμπόριο υψηλής συχνότητας, το layering, για γιατί θα υπάρχουν όλο και νέοι μηχανισμοί και νέα μέσα χειραγώγηση αγοράς, θα πρέπει ίσως μέσω κατεξουσιοδότηση πράξεων να αντιμετωπίσουμε και αυτές τις νέες περιοχές, τους νέους τομείς που αυξάνονται και που αυξάνει η δυνατότητα κατάξυσης αγοράς. Για τις παρεκκλήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρω ότι η Επιτροπή κατ' επανάληψη είπε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα πιο ελαφρύ καθεστώ για αυτέ τι επιχειρήσει. Θα πρέπει να του επιτρέπουμε και να έχουν τα εργαλεία να πληρούν ε, τι προποθέσει τη νομοθεσία. Φυσικά εγώ το θέλω αυτό, αλλά δεν θέλω ε, ελαφρύτερο καθεστώ, το οποίο σημαίνει ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει θα μπορούν και να χειραγωγούν την αγορά και να την γλιτώνουν. Δεν είναι αυτό ο στόχο τη νομοθεσία. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε την σωστή ισορροπία. Δηλαδή, να μην τι βαρύνουμε υπερβολικά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αλλά να μην ανοίξουμε παραθυράκια ε, για χειραγώγηση από τους συμμετέχοντες στην αγορά. Ε, κάποια άλλα θέματα για τις ερευνητικές εξουσίες, ε, άρθρο 17 του κανονισμού, υπάρχει και στην οδηγία MIFID, άρθρο 71, ορισμένες εθνικές αρχές δεν θέλουν να αποδυναμώσουν τη δυνατότητα πρόσβαση δεδομένων ε, σημαντικών για τη δουλειά τους. Ξέρω ότι αυτό το θέμα, Πρόεδρε, ε, θα, το θα το διερευνήσει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Υπάρχει όμως και το διδακτικό της οδηγίας MIFID τη οδηγία μύθη. Θα πρέπει λοιπόν και εμεί να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ορισμένε εθνιστικέ αρχέ πιστεύουν ότι α, η τρέχουσα οδηγία θα του μειώσει τι εξουσίε να ζητούν α, στοιχεία και να τα λαμβάνουν. Θα πρέπει να το δούμε αν όντω έτσι συμβαίνει. Επίση, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Τι κάνουμε με του διευθυντέ που διαπραγματεύονται χρησιμοποιώντας εμπιστευτικές πληροφορίες. Είχαμε περιπτώσει όπου traders ε, σε μια εταιρεία πούμε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, κάποιος ήξερε ε, τα νούμερα διαπραγμάτευσης τα Χριστούγεννα, πούλησε και έβγαλε 300.000 τερλίνες πριν βγει προς τα έξω η πληροφορία. Στον τύπο δεν... αναφέρθηκε ότι δεν διώχθηκε για κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών, γιατί είπε ότι δεν είχε πολύ σημαντικές πληροφορίες αυτό τι σημαίνει, μας επαναφέρει στο θέμα του κατά πόσον έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες οι ρυθμιστικές αρχές. Ένα άλλο θέμα, αν θα πρέπει να έχουμε να δώσουμε δυνατότητα στους διευθυντές ε, να διαπραγματεύονται μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Να έχουν ένα σλότ, ας πούμε. Θα πρέπει να το δούμε με τους stakeholders για να την ψάξουμε αυτή την ιδέα. Αλλά κάπως θα πρέπει να το καλύπτει ο κανονισμός αυτό το θέμα. Επίσης τα αγαθά συμπεριλαμβάνονται και φυσικά ο κλάδος θέλει εξαιρέσεις ή αποδυνάμωση των διατάξεων για τα αγαθά, για το εμπόριο αγαθών. Και η ΜΑΤ και η ΜΥΦΙΔ δεν καλύπτουν το θέμα των αγαθών. Ε, νομίζω ότι τώρα σε αυτή τη νέα νομοθεσία θα πρέπει να καλύψουμε και, την, και τα αγαθά και νομίζω η Κομισιόν το θέλει αυτό. Ε, θα πρέπει να ξαναδώ την οδηγία. Ε, δεν το έψαξα αυτό χωριστά. Θέλω να το καλύψω στις ε, γενικές κυρώσεις. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας γενικός ορισμός, οριζόντιες ας πούμε ποινικέ κυρώσεις. Από ό,τι ξέρουμε από την Κομισιόν, είναι η πρώτη φορά που προτείνονται ποινικέ κυρώσει στον τομέα αυτό. Ε, Ίσως θα πρέπει πρώτα να δούμε την οδηγία πώ δουλεύει στην πράξη πριν την αναθεωρήσουμε, αντί να δημιουργούμε καταλόγους ε, κυρώσεων. Δεν είμαι πολύ πρόθυμη να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θέλω, δεν θέλω να βαρύνω τις ρυθμιστικές αρχές με άπειρους ορισμούς, ας πούμε, ε, πριν τους δοθούν πραγματικά και τα εργαλεία και πριν τα τεστάρουν αυτά τα εργαλεία που θα έχουν στη διάθεσή τους για να ε, δουν πώς θα λειτουργήσει η οδηγία. Επίσης, κυρώσεις για τη συμπεριφορά. Πρέπει να δούμε και αυτό πώς θα λειτουργήσει. Φυσικά δεν πρέπει να είμαστε πολύ επιτακτικοί προς τα κράτη-μέλη. Α το αφήσουμε ως προς αυτό το θέμα ε, κάποια ευελιξία. Νομίζω ότι αρκούν αυτά. Θα δώσω κάποιο χρόνο στους συναδέλφους, στους κοιόδη εισηγητές και ίσως και στην Κομισιόν. Thank you very much. Uh, Mrs. Από όσο γνωρίζω έλαβε στο του... Ε, θα λάβει το λόγο εξ ονόματος τη, του ΕΛΚΑ. Η κυρία μιτιάν δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί εδώ, αλλά θα ήθελα να παρουσιάσω τα δικά της σχόλια. Η βάση παρουσίασης είναι αρκετά καλή. Θα πρέπει όμως να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής έτσι ώστε να ε, υπάρχουν ίσοι όροι πρόσβασης για όλα τα κράτη-μέλη και να ενισχύσουμε και τον κυρωτικό μηχανισμό που προκύπτει από τη χειραγώγηση της αγοράς ή της καταχρήσης. Έχει μεγάλη σημασία Επίσης, η οδηγία MAR να ενταχθεί στο ίδιο χρονικό πλαίσιο με την οδηγία MIFID. Είναι τα δύο πακέτα τα οποία έχουν άμεση συναφία. Εδώ η συγγήτρια έχει θέσει ένα καλό βηματισμό σε σχέση με τον κατακαιρματισμό της αγοράς και τον πολλαπλασιασμό των ε, σημείων συναλλαγής θα πρέπει να βρούμε μία εξισορρόπηση και επίσης να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την, τις καταχρήσεις. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα. Υπάρχει μία ενδιαφέρουσα πρόταση στην ακρόαση MIT έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε το στοιχείο κατακαιρματισμού μέσω του διασυνοριακού, της διασυνοριακής, ε, των διασυνοριακών χρηματιστικών συναλλαγών με βάση τις εισαγωγές στο χρηματιστήριο. Αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο τη βάση συναλλαγής, αλλά θα μπορέσουμε να κρίνουμε και το βαθμό εκτέλεσης και να δούμε ποια ε, προϊόντα ε, έχουν εισαχθεί και τι παραγγελίες έχουν γίνει. Αυτό αφορά την πρωτογενή αγορά και αφορά την, και την προστασία δεδομένων. Και η προστασία δεδομένων θα πρέπει να ενταχθεί στην πρόταση, όμως θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα από αυτού. Γενικότερα, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα σημεία κλειδί του κανονισμού έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα εθνικής ερμηνείας έτσι ώστε να υπάρχουν ίση όροι πρόσβαση σε σχέση όμως με τα άρθρα καθεαυτά του κανονισμού και της οδηγίας θα ήθελα να πω σε σχέση με την, τον ορισμό ως προς τις πληροφορίες εκ των έσω. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η πληροφόρηση είναι συναφής για τους ε, επενδυτές και ότι είναι πληροφόρηση εκ των έσω. Θα πρέπει επίσης να δούμε κατά πόσο οι τιμές που προτείνονται είναι λογικές Όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν στον κανονισμό, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να ειχνηλατήσουμε την κατάχρηση, τις καταχρήσεις αγορές. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ορίσουμε αυτό το θέμα λίγο περισσότερο. Να δώσουμε παραδείγματα δηλαδή, χωρίς ένα διεξοδικό κατάλογο ως προς τους, ε, το συσχετισμό μεταξύ ε, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων και επειδή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το διτό χαρακτήρα θα πρέπει να ξέρουμε ποια αρχή ισχύει και αλλού σε άλλα νομοθετήματα όπου υπάρχουν παρόμοιες διατάξεις για κυρώσεις, δηλαδή στο CRD και στο MIFID. Επίσης, θα πρέπει να μιλήσουμε όχι μόνο για διασυνοριακές περιπτώσεις, αλλά για, το, για εθνικό καθαρά επίπεδο. Αυτά ήθελε να πει η κυρία Κάινεν και θα ήθελε και οι δύο εκθέσεις να βελτιστοποιηθούν κατά το δυνατό. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την Αρλίν για τον τρόπο με τον οποίο μέχρι στιγμής εξέτασε το θέμα, ιδίω νομίζω ότι η ακρόαση που είχαμε στις 24 ε, Ιανουαρίου ήταν πάρα πολύ καλή. Όλοι που συμμετείχαν σε αυτή την ακρόαση συμφώνησαν ότι πρέπει να εξετάσουμε την ελόγω οδηγία γιατί έχουν αρχίσει αρχίσει, ε, έχουν αλλάξει γνώμη οι προϋποθέσεις, η δομή των αγορών είναι διαφορετική, οι εμπορικέ πλατφόρμε είναι διαφορετικές, ο κόσμος διαφορετικό. οι τεχνολογικέ δυνατότητε έχουν προχωρήσει και γι' αυτό πρέπει να έχουμε κάτι το καινούριο. <clears throat> το ενδιαφέρον είναι ότι η Κομισιόν αυτή τη στιγμή προτείνει ένα κανονισμό και μία οδηγία. Το είχαμε ήδη στη Βασιλεία 3 μία φορά. Και αυτό είναι κάτι που δεν χαιρετίζουν ε, ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη που προτιμούν ένα κανονισμό από μια οδηγία. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να εξετάζουμε όσο περισσότερο ε, κανονισμούς γιατί η πρακτική εφαρμογή των επιθυμιών του νομοθέτη έτσι εξασφαλίστηκε στα 27 κράτη-μέλη. Ε, τα περιθώρια λιγμών που πρόσφεραν οι οδηγίες στο παρελθόν δεν θα υπάρχουν πια. Τώρα, συγκεκριμένα σημεία που εν μέρει τα ανέφερε και η Αρλίνη ήδη. το πρόβλημα του πώς θα οριστεί ο λεγόμενος insider, εκείνος που έχει γνώσεις εκ των ένδοα. Η Κομισιόν φαίνεται θέλει να εξετάσει την έννοια αυτή ευρύτερα από ό,τι συνηθίζεται μέχρι στιγμής. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν πολύ ακριβείς κατάλογοι των ατόμων αυτό, πράγμα που σημαίνει συμπληρωματική εργασία. Δεν μπορεί να αποτευχθεί αυτό αποφευχθεί αυτό μας. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι στους οποίους μιλήσαμε θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να το κάνουμε μάλλον. Έχει μια πρακτική αρνητική επίπτωση. Αυτό που προσπαθούμε δηλαδή από την άλλη μεριά όσον αφορά τα συστήματα πληρωμών, οι πληρωμές δηλαδή να εξαρτώνται περισσότερο από τα αποτελέσματα της επιχείρησης υπό τη μορφή ε, μετοχών θα περιοριστεί γιατί ε, αυτός που παίρνει αυτές τι μετοχές είναι insider στην προηγουμένη περίπτωση και αν δεν έχει τη δυνατότητα να τι χρησιμοποιήσει οι μετοχές αυτές όπως θα ήθελε υπάρχει ένα πρόβλημα καθιστά δηλαδή λιγότερο ελκυστική αυτή η προσφορά κατόπιν η αναγκαιότητα να συμβαστούν οι πληροφορίες εκ των έσω και ε, άλλες πληροφορίες που δίνεται. Ένα παράδειγμα σας δώσω. Μία επιχείρηση αποφάσισε να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εξαγοράς των μετοχών της. Έχει ήδη δώσει την εντολή στις τράπεζες να το κάνει αυτό στο χρονικό διάστημα αβ. Τώρα ξαφνικά υπάρχει μια μεγάλη απώλεια της επιχείρησης αυτής γιατί κάποιο εργοστάσιο που ήταν στο εξωτερικό γκρεμίστηκε, δεν ξέρω κάτι τέλος πάντων. Και εκείνη τη χρονική στιγμή αυτή η επιχείρηση δεν θα ήταν σε θέση να διακόψει την εφαρμογή της εντολής που έχει δοθεί και δεν έχει ακόμα εκτελεστεί. Θα έπρεπε δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση το ελεκτικό συμβούλιο αυτή τη επιχειρήση που είναι insider θα πρέπει να αφήσει να λειτουργήσει, να συνεχίσει αυτή η διαδικασία, δηλαδή να επανεξαγοράσει τις μετοχές της εταιρείας, όλο που ξέρει ότι η εταιρεία δεν έχει χρήματα να το κάνει πια. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτές οι, οι περιπτώσεις όπου υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ των γνώσεων των εκ των έσω των insider και των ad hoc αποφάσεων θα πρέπει να εξαστούν καλύτερα. Το επόμενο που αφήνει και η Αρλίν είναι ε, αυτά που κάνουν οι διευθυντές οι λεγόμενοι, οι directors. Θα ήταν πραγματικά καλό να αυξηθεί ο όγκος των ε, συναλλαγών που θα πρέπει να δηλώνονται πολύ περισσότερο από τι 20.000 που προβλέπει η Κομισιόν. Θα ήταν κατά γνώμη μου το ελάχιστο 50, αν όχι και 100.000 που μπορούσα να δεχτώ. αυτό. Το δεύτερο αναφέρεται στην χρονική περίοδο δηλώσεων. Η Κομισιόν λέει αυτή η χρονική περίοδος που είναι 5 μέρες θα πρέπει να μειωθεί στις 2. Εγώ προσωπικά και από την πρακτική εμπειρία που είχα πριν να ξεκινήσω με την πολιτική θα έλεγα ότι αυτή την περίοδο μπορούμε πραγματικά να την ε, μειώσουμε. Τώρα κατά πόσον δύο μέρες είναι υπερβολικά φιλόδοξο δεν ξέρω αυτή τη μεριστικά. Εξεπλάγει όμω που όλοι με τους οποίους συνομίλησα από το θέματος να μου πούνε ότι είναι αδύνατο δύο μέρες. Εγώ το έχω κάνει σε δύο μέρες, δεν είναι δηλαδή αδύνατο τελείω, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ίσως σε ορισμένες χώρες ε, ε, είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι άλλες. Εντάξει, άμα είναι υπερβολικές οι δύο μέρες θα έλεγα ίσως να μην είμαστε τόσο αυστηροί στην ε, μείωση αυτής της ε, προθεσμίας. Αλλά να πληρωθεί είναι. Το τελευταίο σημείο που έχω να παρατηρήσω. Έχουμε βέβαια κάθε συμφέρον να γνωρίζουμε τις ε, ε, καταχρήσεις της αγοράς. Δεν ξέρω όμως εάν το λεγόμενο whistleblowing, η ε, είναι το καλό μέσο. Γιατί κατά κάποιον τρόπο πιέζουμε τους ε, συνεργάτες μιας επιχείρησης να μας δηλώνουν ότι θεωρούν ότι πάει στραβά. Δεν μου φαίνεται ότι είναι πολύ καλή η τακτική αυτή. Το τελευταίο σημείο έχουμε το θέμα των ποινικών κυρώσεων. Δυστυχώ αυτή τη στιγμή σε 27 χρόνια χωρισμένοι υπάρχουν τεράστιε διαφορετικέ. Υπάρχουν χώρε στι οποίε υπάρχει de facto η, η δυνατότητα αστυνομική δίωξη. Σε άλλε χώρε δεν υπάρχει καμία τέτοια δυνατότητα εάν γίνει κάτι γίνεται μόνο λόγω της στενής συνεργασίας της εποπτικής αρχής με τις αστυνομικές αρχές. Και το ότι προσπαθεί εδώ η Κομισιόν να υπάρχει μεγαλύτερη ομοιομορφία είναι οπωσδήποτε αξιόλογο όσον αφορά τους στόχους και καλόδεκτο θα έλεγα. Το θέμα είναι κατά πόσον ε, επί τη ευκαιρία αυτής εδώ της, ε, περίπτωσης να κόψουμε τόσο πολλό τα δικαιώματα της ε, ε, Επικουρικότητα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλέ παρατηρήσει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ελπίζω τι επόμενε εβδομάδε θα μπορέσουμε να διευκρινίσουμε τα πράγματα και προσβλέπω μεγάλο ενδιαφέρον στην έκθεση τη Ελλήν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Πασκάλ. Ή μάλλον. Μάλλον ε, δεν πρόφτασε να έρθει ακόμη ο συνάδελφος κάπου, έχει κολλήσει την κίνηση. Ο Πασκάλ, όπως και προλαλήσατε οι περισσότεροι τουλάχιστον, χαίρομαι και εκ μέρους των Πρασίνων και προσωπικά για την οδηγία και τον κανονισμό που βρίσκονται προς συζήτηση και σε κάποιο βαθμό πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη και πιο φιλόδοξοι. Αλλά παρόλα αυτά και η οδηγία και ο κανονισμός ε, είναι καλές βάσεις εργασίας και μακάρι να έρθουν σε αίσιο πέρας και τα δύο νομοθετικά κείμενα και σε όλες τους τις διαστάσεις. Θα ήθελα να εκφράσω ιδιαίτερα την ικανοποίησή μου και την εναρμόνιση των κυρώσεων. Νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του απολογισμού της πρώτης οδηγίας που ε, έχρισε κατεπηγόντως ε, αναθεώρησης και έχει υποβληθεί στο δεύτερο σχέδιο και η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή είναι δόκιμη. Αυτά θα τα επιδοκιμάσουμε και στη συζήτηση και νομίζω ότι υπάρχει και συνένεση μεταξύ μα, άρα θα δημιουργηθεί και πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά το high frequency trading, τι ε, συναλλαγέ υψηλή συχνότητα, Μερικέ εποπτικέ αρχέ υπέβαλαν ακόμη πιο φιλόδοξε προτάσει από αυτέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ζητώντα, για παράδειγμα να μην ε, καταγράφονται μόνο οι συναλλαγές αλλά και οι παραγγελίες ώστε εκεί να βλέπουμε αν γίνονται κάποιες χειραγωγήσεις κατά χρήση αγοράς μεταξύ των παραγγελιών και των συναλλαγών. Γι' αυτό και θέλουμε να ενισχύσουμε το σημείο αυτού του κειμένου που αφορά το high frequency trading. καλύπτοντας ακόμη και τις παραγγελίες και όχι με περιορισμό τους στις εναλλαγές. Βέβαια το αντεπιχείρημα που υπευλήθη κατά τι πρώτε είναι ότι είναι πολύ δαπανηρή η διεύρυνση του πεδίου και στις παραγγελίες, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν αρκεί το επιχείρημα αυτό, γιατί αν πραγματικά θέλουμε να θεσπίσουμε ένα σύστημα, μπορεί να είναι δαπανηρό, αλλά το να εξασφαλίσουμε τελεσματική υποπτία του και αυτή η άσκηση είναι δαπανηρή, αλλά είναι συνολικό το πακέτο δεν μπορούμε ένα σκέλος μόνο του συστήματος να το χρηματοδοτούμε και το δεύτερο σκέλος στην εποπτεία να τσιγκουνευόμαστε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην εποπτική αρχή. Και αυτή η πληροφορία είναι απαραίτητη, κατά τη γνώμη μου, και οι παραγγελίες. Γιατί το high frequency trading έχει αποκτήσει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις στην αγορά. Φαντάζομαι με τον προλαλήσαντα θα διαφωνήσουμε στο σύστημα προειδοποίησης ε, συναγερμού. Ε, πιστεύουμε ότι ένα σύστημα ε, του συστήματος, ε, το whistleblowers, της προειδοποίησης του συναγερμού, είναι σημαντικό. Βέβαια υπάρχουν και μεμονωμένοι φορείς που ίσως να μην θέλουν να περιληφθούν σε αυτή την διαδικασία και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε προστασία τους αυτούς που κάνουν τις καταγγελίες. Ε, θα πρέπει να προστατεύσουμε τους whistleblowers ε, και να προσθέσουμε κάτι αντίστοιχο στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ό,τι αφορά το trading των, ε, ιδιο, των ιδιοκτησιών, των ιδιοκτητών, συγγνώμη, στις Ηνωμένες Πολιτείες κάποιες τράπεζες ε, φαίνεται ότι θα τους διαφορετική θέση από, αυτές, ε, από τη θέση που συμβούλευαν για τους πελάτες τους. Θα δούμε τώρα τι μέτρα χρειάζονται στην αγορά και τι βαθμός διαφάνειας απαιτείται για να αποφύγουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και για τα σημεία αυτά θα υποβάλουμε προτάσεις πιο φιλόδοξες από τις Ευρωπαϊκές Επιτροπές. Και το τελευταίο σημείο αφορά τις κυρώσεις για τους, ε, καταχρο... τους ε, τους... αυτούς που ε, προβαίνουν στις χειραγωγήσεις. Προτείνονται μερικές φορές οικονομικές κυρώσεις, αλλά παραμένουν στο σύστημα. Και δεδομένου των τεράστιων κονδυλίων και του τζίρου, οι οικονομικές κυρώσεις δεν είναι ιδιαίτερα αποτρεπτικές, μια και κάποιος μπορεί να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Εγώ θα έλεγα να απαγορεύουμε την άσκηση του επαγγέλματος, ορισμένων τουλάχιστον επαγγελμάτων στο χρηματοπιστωτικό κλάδο σε όσους έχουν καταδικαστεί για κατάχρηση αγοράς. Δεν αρκούν οικονομικές κυρώσεις, δεν είναι αρκετά αποτρεπτικές ε, για τους ε, αυτούργους εφόσον θα μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμα. Αυτά είναι κάποια στοιχεία που προτείνουμε για τη βελτίωση του κειμένου. Επαναλαμβάνω ότι η σημερινή εκδοχή και της οδηγίας και του κανονισμού είναι ήδη αρκετά ενδιαφέρουσες. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλους ε, ομίλητες στο κατάλογο, μόνο εγώ έχω απομείνει. Δεν ξέρω αν η Σιλβή θέλει το λόγο τώρα ή μετά. Συμφωνώ. Συμφωνώ με τα περισσότερα σχόλια του Πασκάλ και οι δικές μου σκέψεις για την κατάχρηση αγοράς, όπως είπα, είναι ότι αν τι άλλο, καλύτερα να είμαστε φιλόδοξοι παρά να βάζουμε συνέχεια νερό στο κρασί μας. Στην ακρόαση ακούσαμε κάποιες προτάσεις ότι αφορά την αφιβολία για το επίπεδο της διαστάσης της κατάχρησης αγοράς και μερικοί είπαν ότι ίσως δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα, ίσως δεν γίνεται τόσο σημαντική κατάχρηση αγοράς. Είχαμε όμως και ένα άρθρο στους Financial Times που το κράτησα κιόλα και που ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ότι υπάρχουν κάποιες περίεργες ε, δραστηριότητες στο 1 τρίτο των συγχωνεύσεων. 1 τρίτο δεν μπορεί να κριθεί ε, επουσιώδες ποσοστό. Δείχνει ότι κάτι συμβαίνει και όσο πιο νωρίς εντοπίσουμε τις καταχρήσεις αγοράς, τόσο το καλύτερο. Τώρα αυτό το θέμα των διοικητών, των μετοχών κτλ. είναι αρκετά περίπλοκο εξαιτίας της διαφορετικής φύσης και του χαρακτήρα των επιχειρήσεων. Σε ορισμένες επιχειρήσεις θέλουμε οι διευθυντές να είναι και μέτοχοι, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις. Όταν έχουμε όμως μεγάλες πολυεθνικές οι τράπεζες και ούτω καθεξής, τότε αρχίζουμε και έχουμε κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι δόκιμα ένα τέτοιο μέτριο. Σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις κεφαλαίου, εκεί που έχουμε και τις αμοιβέ, εγώ πάντα προτιμούσα άλλα, άλλα μέτρα κεφαλαίου αντί για μετοχές. Προτιμώ να μην δοθούν κίνητρα ε, να κάνει κανείς ελαθροχειρίες με τις μετοχές του για να αυξήσει την ε, αξία τους. Γιατί εκεί μπορούν να γίνουν διάφορες καταχρήσεις και χειραγωγής αγοράς. Ενώ στα κεφαλογικές απαιτήσει έχουμε αντίστοιχα κριτήρια για να ελέγξουμε το κατά πόσο εφαρμόζονται. Τώρα, έχουμε ήδη μια θεωρία που λέει ότι όταν είναι να αποφασίσουμε κάτι να το σκεφτόμαστε δύο φορές. Αν όμως ε, δεν το κάνουμε καθόλου, τότε έχουμε και ε, αντιπαράθεση με κάποιες ε, ε, διατάξεις που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, του safe harbor που λειτουργούν ως ασφαλής παράδειση κατά κάποιο τρόπο. Γιατί... Ε, ναι, μεν εμποδίζουμε τις καταγγελίες, αλλά όταν έχουμε τις πληροφορίες αυτές από άλλη οδό, θεωρούμε ότι ε, είναι θεμητές. Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε τέτοια παραθυράκια. Ε, και να μην αποθαρρύνονται οι καταγγελίες. Τώρα, μερικές φορές οι καταγγελίες δεν ξέρουμε αν ε, είναι ε, όντως ε, χρήσιμες οι πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά το high frequency trading, δεν είμαι σίγουρη ότι οι αλγόριθμοι ε, ενέχουν αυτό το δυναμικό της χειραγώγησης τους. Πάντως, το θέμα των ακυρώσεων και το γεγονό ότι οι ακυρώσει μπορούν να κρυθούν ω χαρα... Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό μέσω των αλγορίθμων, ίσως με άλλο τρόπο. Πάντως, ο φόρος χρηματοπιστών, ο χρηματοπιστικό συναλλαγών, ακριβώ επειδή φορολογεί και τι ακυρώσει όπως και τις συναλλαγές, ίσως είναι ένα τέτοιο μέτρο. Ίσως είναι ένα καλό τρόπο για να εξασφαλίσουμε το στόχο μας. Αντί να έχουμε τη διάκριση μεταξύ high frequency trading και κανονικού trading. Πάντως, οι ακυρώσει για λόγους χειραγώγησης είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά αν θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητε να, να βρούμε τις ατασταλίες. Αυτά από πλευρά μου, η Σιλβή. Μια παρατήρηση σύντομη και γενική. Θέλω να καλέσω τους εισηγητές και την εισηγήτρια και τους σκιώδη τους Κιώδης, να δουν τι προσπαθήσαμε να, δημιουργήσαμε, να δημιουργήσουμε με την, όταν φτιάξαμε τις εποπτικές αρχές. Τότε είχαμε κάποιους στόχους, μην τους ξεχνάμε. Και όταν συζητήσαμε την ε, ΜΑΔ, συνειδητοποιούμε ότι όταν μπαίνουμε πια στα τομιακά προβλήματα, χάνουμε την ε, συνοδική εικόνα. Ε, όσο περισσότερο είμαστε συνεπείς με αυτά που είπαμε στο παρελθόν, τόσο πιο δυνατοί παραμένουμε. Ακόμα και αν δεν το πετύχουμε αμέσως, θέλουμε έναν έλεγχο στην πραγματικότητα των καταχρήσεων, των κενών, των προβλημάτων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε, χάρη σε μια εποπτεία ευρωπαϊκή και χάρη σε όλα αυτά τα μέτρα που θέλουμε να προωθήσουμε εδώ με αυτά τα νέα νομοθετήματα. Ευχαριστώ. Ωραία. Έχουμε την ε, Κομισιόν, τη Μαρία Τερέζα. Κατάλληλη στιγμή είναι να μπείτε στη συζήτηση για να δώσω μετά το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την επικοδομητική σας συζήτηση, η οποία πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση με την πρόταση της οδηγίας ε, που σκοπό έχει να ενισχύσει το πλαίσιο. Ε, επίσης ε, συνάδει με τις δεσμεύσεις ε, του G20, με τις αρχές de la Rosière. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε αυτή την συνέπεια, ε, να κρατήσουμε τους κανόνες και να τους ενισχύσουμε. Γιατί επειδή πάμε από οδηγία σε κανονισμό, θέλουμε να μην έχουμε δυνατότητα, τα κρατημέ... να μην δώσουμε τα δυνατότητα στα κράτημενα να κάνουν ό,τι θέλουν. Θέλουμε σαφείς ορισμούς. Το είπαν κάποιοι από τους ευρωβουλευτές από της Επιτροπής, ε, ορισμένοι, ορισμένοι δεν είναι ξεκάθαροι. Παραδείγματο χάρη σημαντικέ πληροφορίε. Ε, πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί αυτό ο ορισμό, ούτω ώστε το ε, κείμενο να μην δίνει ε, δυνατότητα έλλειψη ισότιμη μεταχείριση. Για μα στην Κομισιόν το Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη το ΜΥΦΙΤ και το MAD τις ε, δύο αυτές οδηγίες, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ε, φτάσουμε σε μια ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Γι' αυτό έχει σημασία να δούμε τις αρχές, τους στόχους και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Σε σχέση με αυτά που προελέχθησαν, για το διασυνοριακό έλεγχο σημείων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αντιμετωπίσαμε ορισμένα προβλήματα σε σχέση με την διαλειτουργικότητα των συστημάτων ως προς την προστασία των δεδομένων, αλλά δεχόμαστε τις περαιτέρω βελτιώσεις του κειμένου. Θεωρούμε ότι υπάρχουν νομικές δυνατότητες. Επίσης, το θέμα του νέμπις in idem σε σχέση με τις ε, διασυνοριακές καταστάσεις θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ισχύει και σε εθνικό επίπεδο το νέμπις in idem. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να δικαστεί για το ίδιο παράπτωμα δύο φορές. Έχει λοιπόν σημασία να δούμε κατά πόσο στην ε, περίπτωση αυτή δίωξης, κατά πόσο η δίωξη, δηλαδή η δίωξη θα ισχύσει μία φορά. Δηλαδή το nebis in idem αυτή τη φορά έτσι θα πρέπει να ερμηνευτεί ότι θα υπάρξει μία καταδίκη, είτε πρόκειται για ποινική δίωξη είτε όχι. Και γι' αυτό οι αρχές δεν θα πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις δύο φορές με βάση το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προστασία των φυσικών προσώπων. Ως προς τα μέτρα του επίπεδου 2, μας ενδιαφέρει να δούμε πώς αυτή η νέα πλαισίωση θα αντικαταστήσει την τρέχουσα και νομίζω ότι θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή αυτός ο κανονισμός τη στιγμή που θα έχει διευθετηθεί το δεύτερο επίπεδο από την Κομισιόν ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές για να υπάρξει πλήρης αντικατάσταση. Άρα προσμένουμε τη συνέχιση της συζήτησης σε αυτό το θέμα για να φτάσουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα ενισχύσει τον κανονισμό για να προωθήσουμε την προστασία δεδομένων και να δημιουργήσουμε ίσες συνθήκες πρόσβασης προς όλους. Η Αρλίν έχει το λόγο. Ευχαριστώ όλους για τα σχόλια. Πολύ χρήσιμα. Σιλβί, σε διαβεβαιώ ότι στη συζήτηση της τρογγυλής τραπέζης που είχαμε η ΕΣΜΑ ήταν παρούσα, εκπροσωπήθηκε και ακούσαμε α, τις απόψεις της. Θα συνεργαστούμε για το θέμα αυτό της κατάχρησης ε, της αγοράς. Ε, θέλουμε έναν γενικό κανόνα, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι, αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τον πετύχουμε. Κυρία Πετακάνων, το θέμα αυτό έχει τεθεί. Θα το κοιτάξω. Το θέμα του ορισμού της, της εμπιστευτικής πληροφορίας και της σημαντικής πληροφορίας. Επίσης το θέμα της ε, διασυνορικής συνεργασίας και πώς θα έχουμε πρόσβαση σε διασυνοριακές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Ε, δεν είναι εύκολο από Κομισιόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει πρέπει να το κοιτάξουμε. Σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κύριος Κλίντ, χαίρομαι που πιστεύετε ότι θα πρέπει να είμαστε σκληροί στον τομέα αυτό. Αυτό που ήταν πολύ ενδιαφέρον ήταν το αν θα πρέπει να έχουμε κανονισμό ή οδηγία. Οι εθνικές αρχές στο, στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης είπαν ότι ορισμένοι είχαμε ας πούμε την οδηγία μέχρι τώρα και εκείνοι ήταν πολύ πιο αυστηροί, ξεπέρασαν την οδηγία. Γιατί λοιπόν να μην ξεπεράσουμε την οδηγία. Γιατί η οδηγία δεν μας καλύπτει πια όσο πιο πολύ α, εξυγχρονίζονται όσοι κατέχουν εμπιστευτικέ πληροφορίε και χρησιμοποιούν πιο καλέ καλές μεθόδους, πούμε. Το θέμα των εμπιστευτικών πληροφοριών και ποιο τις κατέχει πρέπει να το δούμε. Αυτό που είπατε για τα προγράμματα ε, χορήγησης μετοχών σε διευθυντικά στελέχη, θα πρέπει να το δούμε αυτό χωρίς να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε εταιρείε, ε, η λογοδότηση, η ε, λογοδοσία σε δύο ή σε πέντε μέρες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί να μην μπορούμε να τα καταφέρουμε σε δύο μέρες. Δεν μου αρέσει αυτοί που έρχονται και μου λένε δεν μπορούμε να το καταφέρουμε και τα δεν μου λένε και γιατί. Έχουμε τεχνολογία ε, στη διάθεσή μας και επομένως θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ο στόχο μα να είναι δύο μέρε και όταν τέλο κάποιο δεν τον πετυχαίνει, να μα εξηγεί γιατί δεν τον πετυχαίνει. Τώρα για του καταγγέλλοντε. Ε, συμφωνώ με τον Πασκάλ, πολύ σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Αν κοιτάξετε το άρθρο αυτό στη Financial Times, γιατί η ΕΠΑ είναι τόσο πετυχημένη στην ανείχνευση τη κατάχρηση αγορά, είναι γιατί έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα ε, καταγγελιών. και τους ε, πείθουν αυτούς τους ε, καταγγέλλοντες να καταθέσουν στο δικαστήριο. Ορισμένοι δημοσιογράφοι ε, με ρώτησαν αν έχουμε λιγότερες καταχρήσεις αγοράς ή απλώς αν τους διώκουμε λιγότερο. Απλώς είναι πολύ πιο επιτυχής οι Αμερικανοί και υπάρχει μεγαλύτερη δημοσιότητα γύρω από το θέμα. Παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανείχνευση του προβλήματος οι καταγγέλλοντες. Δεν νομίζω ότι με την οδηγία περί ποινικών κυρώσεων θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στην επικουρικότητα. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε ποινικέ κυρώσει. Αν κοιτάξετε το παράδειγμα των Αμερικανών, που επιτρέπει ορισμένα πράγματα στο Υπουργείο δικαιοσύνη, είναι να επισύσει την απειλή αυτή, ότι θα διωχθεί, ότι θα μπει στη φυλακή κτλ. Έχουν όμως και τα DPA που είναι ε, συμφωνίες με την εισαγγελία. Που λέμε ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν θα σε διώξουμε ποινικά, αλλά θα σου επιβάλλουμε ένα πολύ ψηλό πρόστιμο και στις τελευταίες 23 υποθέσεις ε, διώξεων ε, τελικά επιβάλλαν πρόστιμα, δεν προέβησαν στην ε, ποινική δίωξη και κέρδισε το Υπουργείο Δικαιοσύνης 2,3 δις δολάρια. Φυσικά εμεί δεν έχουμε τέτοιο Υπουργείο δικαιοσύνη που θα μπορούσε διασυνοριακά να επιτύχουν κάτι τέτοιο, αλλά θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε στις ρυθμιστικέ αρχές έτσι ένα εύρο, μια ευελιξία, ας πούμε, να χρησιμοποιούν αυτές τις κυρώσει. Παραδείγματο χάρη στην ε, Γερμανία, α, το συνταγματικό δικαστήριο θα πρέπει να δει α, την νομοθεσία που θα επιβληθεί εθνικά για την εφαρμογή για τη μεταφορά τη νομοθεσ... Νομοθεσία ευρωπαϊκής στη Γερμανία. Επομένω δεν πρέπει να είμαστε πολύ επιτακτικοί, πολύ λεπτομερεί ε, ως προς τις ρυθμιστικέ αρχές. Για το πέρασμα από τις 20-50 ή 100.000 λέει ο κύριος Κλίντ. Τι θα γίνει με το κατόφλι. Θα το κοιτάξω. Αν πρέπει να ανέβει στα 50, στις 50.000, στις 100.000 ε, κτλ. Αν έχετε ιδέες, πέστε μου κι εσείς, λέει η κυρία Μακάρθη. Εγώ δεν ήθελα να σας πω ότι δεν θα είσαστε συνεπείς ε, και ότι η δουλειά που κάνουμε εδώ δεν έχει συνέπεια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω στη συζήτηση που θα γίνουν ε, τον, ε, του, τριμερούς, του τριμερή διαλόγου, τριμερούς διαλόγου μάλλον, είναι τα κράτη-μέλη να έχουν συνέπεια, λέει και στην τελική φάση που είναι ο τριμερή διάλογο, τα κράτη-μέλη να έχουν συνέπεια με αυτά που είχαν δεσμευ... συμφωνήσει χρόνια πριν, το 2010 α πούμε. Σα εμπιστεύομαι και σα ενθαρρύνω να εξασφαλίσετε αυτή τη συνέπεια. Υπάρχει μια ερώτηση, δεν ξέρω αν η Αγγλίνη Κομισιόν μπορεί να την απαντήσει. Για αυτή την αναβολή της δίωξης στις ΗΠΑ. Αν θέλουμε να κρατήσουμε και αυτό το ενδεχόμενο ανοιχτό, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ότι γιατί αυτή η επιλογή μεταξύ διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων δεν θα πρέπει να μας ε, δημιουργήσει ε, φραγμούς και τροχοπέδες. Χρειαζόμαστε, λέει η κυρία Μακάρθη, και τα δύο. Ε, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, ευέλικτοι ούτως ώστε να ξέρουμε, να βλέπουμε σε κάθε περίπτωση τι θα χρησιμοποιήσουμε. Ούτε στην Αμερική το προδικάζουν αυτό. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Έχω εδώ ένα προσχέδιο χρονοδιαγράμματο που εξαρτάται βέβαια από το πότε θα υποβάλει η συγκέντρια την έκθεσή Αλλά εγώ βλέπω θα πρέπει να το συζητήσουμε στις 26 Μαρτίου με προθεσμία 24 Απριλίου για τι τροπολογίε και να το εξετάσουμε στι 13 Μαΐου και να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μα τον Ιούλιο με στόχο ενδεχομένω την Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. αλλά ελπίζω να το ζητήσουμε πραγματικά σε 16 Μαΐου. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επόμενο θέμα σήμερα σε διάταξη είναι η δημόσια ακρόαση σχετικά με την πρόοδο επιβολή φόρου και χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ που προβλέπεται στι 5. Δεν έχει ειδοποιηθεί κανένα να έρθει νωρί, άρα έχουμε μισή ώρα διάλειμμα πρωτού μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Εκτός ε, αν κάποιος θέλει να πει κάτι άλλο. Εγώ θα έλεγα να έχουμε ένα διάλειμμα μισή ώρα. Buenas tardes, κυρίες και κύριοι. Θα συνεχίσουμε το εξή θέμα της ημερήσιας διάταξης. Θα συνεχίσουμε με την ακρόαση, τη δημόσια ακρόαση για την πρόβαση, ε, πρόταση επιβολής φόρου στις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές μέσα στα πλαίσια της ε, πρότασης της Κομισιόν για έναν φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Στόχος αυτής της συζήτησης είναι να ορίσουμε την ενδεχόμενη βάση αυτού του φόρου, καθώς και το ποσοστό αυτού του φόρου, την ποσοστία του αναλογία και να δούμε ποιοι θα ήταν οι φορείς ή τα πρόσωπα που θα κατέβαλαν αυτό το φόρο. Επίσης, θα συζητήσουμε για τον ε, τρόπο ε, ίσπραξης αυτού του φόρου καθώς και θα αναλύσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις, τις χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις που θα είχε η εισαγωγή αυτού του φόρου. Όπως γνωρίζετε, έχουμε τέσσερις ε, εισηγητές. Ο καθένας ή η καθεμία θα μιλήσει για 7 λεπτά και μετά θα αρχίσει μία συζήτηση και θα φτάσουμε και στα ε, συμπεράσματα της εισηγήτριας της κυρίας Ποδηματά. Δίνω το λόγο στον κύριο Φίνας Φερσότ που είναι ο πρόεδρος της Intelligence Capital. Έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Good afternoon. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καταρχήν το ιστορικό υπόβαθρο των παρατηρήσεών μου ε, είναι το εξής. Τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας μου ήμουν ε, στην ε, Morgan, UPS, State Street και άλλες τράπεζες ως διοικητικός ε, σύμβουλος. Σε ό,τι αφορά την, το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ακούσαμε επιχειρήματα των πολεμίων του φόρου και θεωρούμε ότι είναι ανεδαφικά τα επιχειρήματα αυτά με βάση την ε, σταδιοδρομία που είχα. Οι Κασάνδρες μπορεί να κραυγάζουν ότι ένας ευρωπαϊκός φόρος χρηματοπιστών συναλλαγών είναι ακόμη μια παλαβή ιδέα των Ευρωπαίων ηγετών που θα προμηνήσει ένα χρηματοπιστωτικό αρμαγεδόνα ε, μερικές φορές επιχειρηματολογούν αυτές οι κατα... κασάνδρες ότι θα καταστρέψει την ρευστότητα θα καταστρέψει τους φορολογούμενους, όχι τους ε, τραπεζικούς και θα εμποδίσει μια ήδη ευάλωτη οικονομική ανάκαμψη. Στην ουσία ο φόρος αυτός είναι πολύ πιο εφικτός από ό,τι θα φανταζόμασταν πολύ. Και όπως και όλοι οι φόροι μπορεί να θεσπιστεί με σωστό ή λάθος τρόπο. Και αν θεσπιστεί με σωστό τρόπο και ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μπορεί να αποφέρει πολλά ωφέλη. Η πολέμη του φόρου αυτού θα ήθελα να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι οι υπέρμαχοι του φόρου είναι παράλογοι, απρεπείς και ε, είναι χρήσιμο να θυμόμαστε ότι ο φόρος αυτός έχει πολύ, μια πρώτη τάξη καταγωγή. Στον αγγλοσακονικό κόσμο, ο Τζον Μέιναρτ Κέιν στον πρώτο ε, ε, πρότεινε στη γενική θεωρία του και μάλιστα ο νομπελίστας James Tobin ακολούθησε το 1971 μέσω της ε, καταστροφής του συστήματος του Bretton Woods. Και το 2009 ο πρόεδρος ε, της Βρετανικής Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, ο Λόρδος Αντέα Τένερ, ε, άφησε κατάπληκτους τους τραπεζικούς του Λονδίνου, κρίνοντας ως σωστή ιδέα αυτό το φόρο. Μεταξύ αυτών των προτάσεων, Μερικοί τραπεζικοί και πολιτικοί προσπαθούν να ξεπλύνουν την κοινωνική του συνείδηση, λέγοντας ότι ο φόρο οπτικό συναλλαγών στη θεωρία είναι καταπληκτική ιδέα, αλλά στην πράξη ανέφικτο. Οι χρηματοπιστές αγορές είπαν ότι περάσαμε από τους ίδιους ελέγχους ε, σε συναλλαγές με φυσική παρουσία, με ταινίε ε, με κωδικούς μετοχής και γραπτές παραγγελίες στον κυβερνοχώρο, που με κανένα δύο κλικ ο επενδυτής χρηματιστηρίου μπορεί να παραπευθεί στο χρηματοπιστωτικό κέντρο με το χαμηλότερο κόστος ε, των συναλλαγών, φόρων και κανονισμών. Είναι πολύ καλή αυτή η εικόνα και γνωρίζω καλά το επιχείρημα γιατί και εγώ το χρησιμοποίησα. Βέβαια, παρά τη λογική αυτή και όλος παραδόξως ε, παρά τη λογική της συνεχούς απάντησης της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου ότι θα υποστηρίξει ένα φόρο μόνο όταν είναι παγκόσμιος για να αποφευθεί η φοροαποφυγή και για να περιοριστεί η φοροαποφυγή, στην ουσία είναι ένας από τους παλαιότερους και μεγαλύτερους φόρους χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ε, λειτουργεί επιτυχημένα και μάλιστα από μόνος του, χωρίς να εφαρμόζεται παγκοσμίω σε ένα από τα μεγαλύτερα ε, και διεθνή, και πιο αθυρά διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα του κόσμου, το Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 1986 και προηγουμένω σε άλλε περιπτώσεις, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου μόνο μερός και χωρίς να περιμένει μιμητές, εφάρμοσε ένα τέλος χαρτοσύμου ε, με συντελεστή 0,5% στις συναλλαγές του Ηνωμένου Βασίλειου, σε μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Και παρόλο που δεν τον επικαιροποίησε προκειμένου να λάβει υπόψη κάποια παράγωγα ή να το επεκτείνει σε αγορές ομολόγων, να λάβει υπόψη και άλλα καινοτόμα προϊόντα ή να μειώσει το συντελεστή προκειμένου να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του χρηματοπιστικού συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, ο φόρος αυτός εξακολουθεί να εισπράττει ετησίως 5 δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής. Βέβαια, Έχουμε και τον φόρο του 0,50% της Σουηδίας που δεν λειτουργήσε σε αντίθεση με τον ε, Βρετανικό φόρο και μάλιστα ο λόγος που λειτουργήσε ο χώρος αυτός είναι ότι είναι ένα τέλος ε, χαρτοσύμου για τη μεταβίβαση κυριότητας. Δεν στηρίζεται στη φορολογική έδρα. Και ε, μπορεί κανείς να μεταβιβάσει κυριότητα σε έναν τίτλο που δεν θα είναι νομότυπος αν δεν έχει καταβληθεί αυτό το τέλος χαρτοσύμου. Δεν θα μπορέσει δηλαδή η μεταβίβαση να εκτελεστεί νομικά σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί αυτό το τέλος χαρτοσύμου. Και μάλιστα οι περισσότεροι ε, δεν αναλαμβάνουν κινδύνους ό,τι αφορά την ε, νομική εκτελεστότητα και μάλιστα 40% ε, ε, των φόρων αυτών καταβάλλονται από ε, ε, κατοίκους στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και μάλιστα πολύ περισσότεροι αλλοδαποί πληρώνουν αυτό το φόρο από οποιουσδήποτε, αντί να οδηγήσει σε έξοδο των φορολογουμένων. Και μάλιστα το Λονδίνο δεν είναι το μόνο αθυρό χρηματοπιστωτικό κέντρο με τέτοιο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Από τις πιο δυναμικές ε, περιοχές και κέντρα χρηματοπιστωτικών στον κόσμο έχουν τέτοιους φόρους χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Η Βομβάη, για παράδειγμα, το Χονγκ Κόνγκ, η Σεούλ, το Johannesburg, η Ταϊπέη έχουν τέτοιου φόρους και από κοινού αυτά τα χρηματοπιστωτικά κέντρα εισπράττουν 23 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Δεν είναι καμία θεωρία, δεν είναι καμία υπόσχεση. Κάθε χρόνο τα κέντρα αυτά συλλέγουν 23 δισεκατομμύρια δολάρια και μάλιστα δεν περιλαμβάνονται εκεί τα τέλη που εισπράττουν clearing houses σε ψηφιστικά γραφεία και ρυθμιστικές αρχές όπως ένα αντίστοιχο που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλοι οι φόροι αυτοί είναι κίνητρα για φοροαποφυγή. Ε, πέραν τη νομική εκτελεστότητα, ένα σωστό φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα πρέπει να είναι χαμηλό, στο μέγεθος, ε, μέτριος, αν, αντίστοιχα με το κόστος των ε, συναλλαγών και να καλύψω στο δυνατό περισσότερους μηχανισμούς αντικατάστασης όσο γίνεται. Και μάλιστα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει ε, την πρότασή της, κάνοντας την πιο απλή, αντί να περιλαμβάνει πολύ περισσότερα εργαλεία οι τράπεζες άρχισαν να υποβάλουν και το υποβλητικό επιχείρημα της ρευστότητα, πολλό δε μάλλον μετά την κρίση που είχαμε το 2008. το βασικό θύμα των φόρων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι αυτοί που ασχολούνται με trading υψηλή συχνότητα. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συνταξιδοτικά ταμεία, ασφαλιστικέ επιχειρήσει και μεμονωμένου επενδυτέ που αλλάζουν πολύ πιο σπάνια το χαρτοφυλάκιό του. Και μάλιστα η μέση περίοδος ε, ε, κράτησης μιας μετοχής ε, ενός συνταξιδοτικού ταμείου είναι δύο χρόνια. Οπότε ένας φόρος χρηματοπιστωτικός αναλόγου για την αγορά αυτής της μετοχής θα πληρώνεται κάθε δύο χρόνια. Φαίνεται βέβαια ότι οι τραπεζικοί θα μετακυλήσουν το φόρο στους πελάτες τους. Αλλά το μεγαλύτερο τμήμα του φόρου δεν θα πληρωθεί από τους φορολογουμένους ή τους συνταξιούχους, αλλά από τους ε, επενδυτές υψηλής συχνότητας. Και μάλιστα επειδή ε, τα hedge funds περιορίζονται σε συγκεκριμένους επενδυτές, είναι και πολύ προοδευτικός αυτός το φόρος. Βέβαια οι high frequency traders λένε ότι αυτοί ε, συνεισφέρουν στη ρευστότητα της αγοράς. Είναι παραπλανητικό όμως αυτό το επιχείρημα. Είχαμε βέβαια ε, αγορές πολύ ρευστές και πριν την εμφάνιση αυτών των ε, ε, επενδυτών υψηλής τυχνότητας. Και μάλιστα σε περιπτώσεις αγοράς με μεγάλη ρευστότητα την υποστηρίζουν οι high frequency trades traders. Αλλά σε περίπτωση κρίσης οι traders αυτοί προσπαθούν να στραγγίσουν την ρευστότητα και μάλιστα σε μια εποχή που χρειάζεται πολύ περισσότερο. Όπως είδαμε στο κράχα στραπής της Νέας Υόρκης της 6ης Μαΐου του 2010. Αν λοιπόν αυτή αυτός ο φόρος χρηματοστικών συναλλαγών να ε, μειώσει το trading υψηλή συχνότητα, μπορεί να, ε, να βελτιώσει την αντοχή του συστήματος γενικώ. Σας ευχαριστώ. Για 7 λεπτά τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σόνι Καπούρ που είναι ο εκτελεστικός διευθυντής του Think Tank Redefine. Έχετε το λόγο παρακαλώ για 7 λεπτά. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το να μιλάει κανένα μεταναστή είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν έχει πια τα επιχείρηματα που χρειάζονται ε, θα προσπαθήσω πάντω. Ποιοι είναι οι στόχοι αυτή τη συζήτηση για τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα που έχουν ακουστεί. Ο ένα λόγο είναι να συλλεχθεί εισόδημα από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, να έχει δηλαδή μια δίκαια συμβολή και ο τομέα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει γενικά σφαιρικά έλλειμμα εισοδήματό ιδίω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με με τραλιτότητε που μπορούμε εκεί να συμβάλλουμε για να χρηματοδοτούν ε, δημόσιες αγορές, ε, κλιματολογικές αλλαγές κλπ. Μετά υπάρχει το επιχείρημα που λέει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η λειτουργία των χρηματοδοτών αγορών και το τέταρτο ότι θα ελιστοποιηθεί η πιθανότητα χρηματοδοτικών κρίσεων. Αυτή η στόχη, όσο και αν είναι ελκυστική, ε, δεν ξέρω κατά πόσον μπορούν πραγματικά να συμβιλιοστούν με έναν φόρο. Αυτός ο φόρος ποια μορφή θα μπορεί να έχει και πώς θα διέφερε η πραγματική μορφή από την πρόταση αγοράς της ε, Κομισιόν. Ε, είναι καλή η πρόταση Κομισιόν όσον αφορά το εύρος που καλύπτει. Όσον αφορά την πρόταση των ε, πολιτών που αναφέρει η Κομισιόν, εάν κανένας σκέφτεται παγκόσμια, ίσως είναι καλό το επιχείρημα ίσως λειτουργήσει και αρκετά αποτελεσματικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όσο πιο ευρέως πρόκειται να εφαρμοστεί ο, φόρος αυτός, τόσο λιγότερο αποτελεσματικός είναι. Σε εθνικό επίπεδο, λόγω του περιορισμένου πολιτικού, της περιορισμένης πολιτικής βούλησης που υπάρχει σε πολλές χώρες υπέρ του το φόρου αυτού, ε, επειδή και μία από τις 27 θα μπορούσε να επιβάλλει βέτο και να οδηγήσει σε καταστροφή της ιδέας αυτής, ίσως υπάρχει κάποιο λογικό όπως ε, το ε, τέλος χαρτοσύμου που λέει για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Αυτή είναι μια αρχή που ισχύει στην αγορά γενικά. Κάθε temptor. Πρέπει να ο αγοραστής να είναι προσεκτικός. Αν αγοράσει κανένα εκλεμμένο αυτοκίνητο, ε, ο τίτλος του αυτοκίνητου, κατοχής του αυτοκίνητου που έχει, έχει μόνη αξία εάν είχε αξία αυτός που τον πούλησε. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Εάν πραγματικά κάποιο αγοράσει ε, μια μετοχή από ένα hedge fund στην ίσως του Καϊμάν, όπου δεν ξέρω κατά πόσο έχει πληρωθεί μια ε, ένα τέτοιο φόρο των συναλλαγών είναι λίγο πιο ακριβή η συναλλαγή αυτή από ότι ε, σε άλλες επιχειρήσεις που ξέρουμε ότι έχουν πληρώσει το φόρο. Ο κίνδυνος όμως είναι τόσο μεγάλος ότι θα χάσω τα χρήματα που έχω καταβάλει που δεν θα το έκανα ποτέ. Ακόμα και αν η Κομισιόν το Κοινοβούλιο που αποφασίσει να προχωρήσει με την αρχή αυτή των κατοίκων θα πρέπει να είναι συμπληρωματική αρχή. Όσον αφορά το θέμα των εξαιρέσεων του μεσάζοντες. Η, η πρόταση της Κομισιόν δεν προβλέπει αυτή την εξαίρεση. Πολλές φορές ακούει κανένας και το χρησιμοποιήσει αυτό το επιχείρημα πως ε, ο φόρος τέλου χαρτοσύμου στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργεί καλά. Όμως είναι ένας φόρος που δεν είναι καλά ε, δομημένος γιατί πλήττει τους τελικούς χρήστες και εξαιρεί τους μεσάζοντες. Το θα ήταν πολύ καλύτερο, θα ήταν χαμηλότερο επίπεδο φόρου που επιβάλλεται σε όλους και στους μεσάζοντες. Γιατί οι high frequency ε, players, ε, οι έμορφη υψηλή συχνότητα δεν πληρώνουν αυτή τη στιγμή αυτό το τέλο στον Βασίλειο. Το πληρώνουν όμω συνταξιούχοι. Και αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί. Το πιο σημαντικό τμήμα τη πρόταση της Κομισιόν είναι ότι η σημερινή προσέγγιση είναι κάπω άχρωμη. Δεν λαμβάνει υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικών τύπων προσωπικέ αγορέ που λειτουργούν διαφορετικά. Η οικονομική το οικονομικό περιεχόμενο δηλαδή, των συναλλαγών είναι διαφορετικό και ο, διαφορετικές αγορές θα πρέπει να έχουν διαφορετικά ποσοστά. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η σημερινή προσέγγιση έχει σαν κύριο στόχο τη δημιουργία εισοδήματο. Αυτό που συστήνουμε εμεί είναι μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση στου φόρου χρηματοπιστικών συναλλαγών, όπου θα υπάρχει καταρχήν προσοχή στην διακανοστική δυνατότητα των φόρων αφών, ε, αυτών, μειώνοντας το συστηματικό κίνδυνο. Το αποτέλεσμα θα είναι τελικά ότι θα υπάρχει κάποιος ισο, ε, κάποιο εισόδημα. Δηλαδή, η ιδέα είναι, εάν υπάρχουν δύο διαφορετικών ειδών συναλλαγών, υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ε, των συναλλαγών over the counter, γιατί αυτές συμβάλλουν περισσότερο στο συστημικό ε, κίνδυνο. και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν και διαφοροποιημένα ποσοστά του φόρου ή παραδείγματος χάρη οι αγορές μετοχών και οι αγορές ομολόγων. Στις ε, αγορές ομολόγων υπάρχει διαφορά ε, ανάλογα με το πότε καθιστώνται με τα ομόλογα αυτά. Και θα πρέπει να εφαρμοστεί ο φόρος ανάλογα. Τα swap μπορούν να αφορολογηθούν βάσει του λεγόμενου delta, δηλαδή θα πρέπει να δούμε πώς διαφοροποιείται η τιμή των ε, παραγόγων από ανάλογα με τον τύπο αυτόν. Εγώ θα υποβάλω ε, μια επίσημη πρόταση στο Κοινοβούλιο με όλες τις λεπτομέρειες της πρότασής μου εξ της ε, ομάδας που εκπροσωπώ, του Redefine. Δεν θέλω να κάνω τώρα κάποιε παρατηρήσει όσον αφορά τι επικρίσει που έχουν ακουστεί για τον φόρο νομοσωπικών συναλλαγών. Η ανάπτυξη θα πληγεί σημαντικά. Η σωστή ερώτηση δεν είναι κατά πόσον εάν αυξηθεί η φορολογία με 15 δισεκατομμύρια ευρώ θα πλήξει την ανάπτυξη ή όχι. Το θέμα είναι ποιος είναι ο λιγότερος φιλικός προς την ανάπτυξη τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα για να εισπράχθουν 15 δισεκατομμύρια. Και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι η απάντηση σε αυτή τη δεύτερη ερώτηση είναι η αύξηση των ε, ε, φόρων χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών, όχι άλλων φόρων. Επίσης, όταν αναφέρονται οι επικρίσεις του τέλους χρωστοσύμου κλπ. Έχουν να πω ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αγορές αυτές δεν συμβάλλουν στην δημιουργία κεφαλαίου. Δεν χρησιμοποιούν οι εταιρείε ε, ε, τα χρηματιστήρια για να αυξήσουν τα κεφαλαιά τους. Ίσως θα υπάρχει υψηλότερο ποσοστό χρήσης των δανείων από τις επιχειρήσεις. Δηλαδή οι επιπτώσεις στο κόστος του κεφαλαίου είναι σχετικά μικρό, μικρές. Και μετά, όσον αφορά τους, ε, τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας. Η ιδέα ότι οι άνθρωποι αυτοί συμβάλλουν στη ρευστότητα και οδηγούν σε μεγαλύτερη ασφάλεια είναι μία από τις πιο επικίνδυνες ιδέες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα η ρευστότητα προέρχεται από πολλού ε, παίχτες τη αγορά. Εάν έχετε μια αγορά στην οποία 70-80% των συναλλαγών γίνονται από ανθρώπου που δρούν κατά τον ίδιο τρόπο, μειώνουν τη διαφοροποίηση και τη ρευστότητα τη αγορά. Και ίσως η κάθε συναλλαγή είναι φθηνότερη, αλλά κάνουν πολύ περισσότερε συναλλαγέ και πληρώνουν συνολικά πολύ περισσότερο. Ευχαριστώ κύριε Κάπο, ο πρόεδρος. Griffith Jones ε, ε, από την Columbia University, διευθυντής του, του προγράμματος που, τον ακολουθεί, που τα ακολουθεί. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να μπορώ να σας προσφωνήσω για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Για το φόρο χρηματοπιστωτικών αλλαγών έφτασε πια ο χρόνος εφαρμογής αυτού του φόρου. Ε, έχει συζητηθεί εδώ και δεκαετίες, όπως είπε και ο Άβινας Περσό, ε, προήλθε από τον Κέινς αλλά ε, είναι συναφής σήμερα μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής κρίσης. Καταρχήν, θα οδηγούσε σε αύξηση φορολογικών εσόδων τη στιγμή σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν υψηλά ε, χρέη και ελλείμματα. Ο φόρος αυτός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μερικός ή ολοκληρωτικός για την δημοσιονομική εξυγίαση που είναι ένας ευκταίος στόχος, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλοί άλλοι. Θα μειώσει το κόστος δανεισμού για τις κυβερνήσεις, καθώς και τη δρυμύτητα των ε, κρατικών χρεών. Επίσης, ε, μειώνοντας ε, το, τα ελλείμματα, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στη συσσόρευση του κεφαλαίου από τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, ένας άλλος παράγων εφαρμογής του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα ήταν να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία, να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις και να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση του πλανήτη, δηλαδή να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Επίσης θα βοηθούσε τις κυβερνήσεις, τη χρηματοδότηση, επενδύσεων για τις πράσινες υποδομές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα αποτελούσε καταλήτη για το, τις αυξανόμενες επενδύσεις και καινοτομία των ΜΜΕ. Επίσης θα είχε μεγάλη ε, σημασία για τη συνολική ζήτηση και τη συνολική προμήθεια. Εάν χρησιμοποιηθούν έστω και έμεσα αυτά τα μέσα, δηλαδή για την ανακεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ, οι επιπτώσεις μόχλευσης θα είχαν ακόμα μεγαλύτερη επίπτωση στην ανάπτυξη. Άρα αυτή η μεγαλύτερη επένδυση, δανειοδότηση θα βοηθούσε στην ανάπτυξη. Εάν λάβουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει μεγάλη ζήτηση και έχει επίσης πολύ περιορισμένη πρόσβαση στη, στη δανειοδότηση. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και από την ε, έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα είχε βαθμιαία εφαρμογή. Και αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα των ε, νοικοκυριών θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν γιατί τα νοικοκυριά θα μπορούσαν να δαπανίσουν ένα υψηλότερο ποσοστό του εισοδήματός τους. Και αυτό αφορά και σχετικότερα πιο ε, πλούσια νοικοκυριά. Αν λοιπόν ισχύσει αυτός ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της και μόνο λίγοι θα καταβάλουν το κόστος, όπως οι ε, χρηματιστές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για έναν πολύ ε, σημαντικό τομέα, δηλαδή πρόκειται για ένα πολύ μικρό μέρος της κοινωνίας με πολύ μεγάλη επιρροή. Ε, βεβαίως ελέγχθη ότι ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα ήταν πολύ κακός για την ρευστότητα, για την ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο. Ε, εσείς ζητήσατε να το συζητήσουμε. Εμείς κάναμε ορισμένες ε, εκτιμήσεις και θεωρήσαμε ότι ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα αυξήσει το ΑΕΠ και θα έχει και όλους ε, του, όλες τις θετικές επιπτώσεις που προανέφερα. Μιλάμε για απώλεια ΑΕΠ της τάξης του 0,50%. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε αυτό το πρότυπο και όπως είπε και ο Σόνι Καπούρ, μόνο το 50% ε, των επενδύσεων θα χρηματοδοτείται μέσω αυτού του φόρου, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ιδιωτικός τομέας χρηματοδοτείται από τα δάνεια των τραπεζών. Άρα μιλάμε για ένα 15% της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Και αυτό αφορά και τις κινητές αξίες οφειλών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν ότι η αρνητική επίπτωση θα ήταν πολύ χαμηλότερη. Μάλλον με συγχωρείτε, η Επιτροπή κρίνει ότι η επιπτώση θα ήταν της τάξης του, 0, του μείον 0,2%. Επίσης υπάρχουν και άλλοι παράγοντες Μιλάμε για την μείωση των συναλλαγών υψηλής συχνότητας που αποτελεί ένα πολύ υψηλό ποσοστό των συναλλαγών και δεν θα είχε αρνητικές επιπτώσεις. Με τον Άβυνας θεωρούμε ότι θα υπήρχαν θετικές επιπτώσεις διότι οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας μπορούν να αποσταθεροποιήσουν την αγορά. Άρα θεωρούμε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις θα ήταν της τάξης του μείον 0,1%. Όμως, αυτές οι εκτιμήσεις, όσο καλές και να είναι, δεν λαμβάνουν υπόψη έναν βασικό παράγοντα, ότι δηλαδή ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα μειώσει τον συστημικό κίνδυνο. Δηλαδή δεν θα είχαμε τόσο υψηλό κίνδυνο να ανακύψουν άλλες χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει και μία χρηματοοικονομική εποπτεία. Αλλά επειδή ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα μειώσει τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας, θα αποθαρρύνει και τις μελλοντικές κρίσεις. Γνωρίζουμε από μελέτες των Reinhardt και Rogoff ότι μετά από κάθε κρίση το ΑΕΠ πέφτει τουλάχιστον κατά 7%. Ε, αν το δούμε αυτό συντηρητικά και δούμε ότι ο φόρος αυτός θα μειώσει τις μελλοντικές κρίσεις κατά 5% τότε θα υπήρχε μία μελλοντική επίπτωση της τάξης του συν 2,5%. Και αν ε, συγκρίνουμε και τον τομέα του, τον ιδιωτικό τομέα, των ιδιωτικών επενδύσεων δηλαδή, θα βλέπαμε ότι θα είχαμε ακόμα ένα μεγαλύτερο ευεργέτημα, κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Αλλά όπως είπε και ο James Tobin, θα πρέπει να δούμε τις θετικές επιπτώσεις. Δηλαδή, ένα, εάν ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μειώσει τα έσοδα του χρηματοοικονομικού τομέα κατά ένα μικρό ποσοστό, και μειώσει τα, τις υψηλές, ε, τα υψηλά έσοδα των ε, χρηματιστών, τότε τα πιο λαμπρά μυαλά θα ασχοληθούν με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, θα πούν στην έρευνα, στην καινοτομία και θα βοηθούσαν για την ε, μελλοντική ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. Έχετε 30 δευτερόλεπτα μόνο. ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν θα συνεισφέρει μόνο στην ανάπτυξη, αλλά στην καλύτερη ανάπτυξη, πιο δίκαιη ανάπτυξη που είναι ύψης της σημασίας τη στιγμή που υπάρχει άνηση κατανομή εισόδημάτων και θα ήταν και πιο βιώσιμη η ανάπτυξη. Γιατί εάν μιλάμε για, πράσινη, για πράσινες επενδύσεις και τις προωθήσουμε, τότε θα ήταν πιο ε, αποδοτική. Ο κύριος Ρίτσαρντ Ρέμπον έχει το λόγο. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εταιρικών Ταμείων. Έχετε 7 λεπτά. Μόνο παρακαλώ. Σας παρακαλώ σεβαστείτε το χρονικό διάστημα που σας δίνουμε. Άκουσα τους τρεις ομιλητές ε, και μετά από αυτό σκέφτηκα να σκίσω την ομιλία μου, θα το κάνω. Σας ευχαριστώ που με καλήσατε. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συμπεριλαμβάνει ε, ταμείες από εταιρείες από 17 κρατημέλη, τη Σουηδία και την Κροατία. Δεν, είμαστε, δεν πιέζουμε υπέρ μεμονωμένων τομέων και δεν έχουμε κανένα κέρδος, ούτε έχουμε εμπορικό κίνητρο πέρα από το βασικό μα σκοπό που είναι να υποστηρίξουμε την επαγγελματική ανάπτυξη όσου δουλεύουν στα ταμεία των επιχειρήσεων, είμαστε και η φωνή των τελικών χρηστών των χρηματοπιστωτικών συστημάτων από την πραγματική οικονομία. Τα άτομα τα οποία δουλεύουν στα ταμεία και σε αυτέ τι ενώσει είναι ουσιαστικά άτομα τα οποία δουλεύουν για κατασκευαστικές ε, βιομηχανίες και για εταιρείε παροχής υπηρεσιών. Βασική τους δραστηριότητα είναι να διαχειριστούν τον επιχειρηματικό κίνδυνο και να εξασφαλίσουν την ρευστότητα και τη χρηματοδότηση, ούτως ώστε να υποστηριχθεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Ο κίνδυνος ε, τον διαχειρίζονται με τα παράγωγα. Δεν θέλουν ούτε να κερδοσκοπήσουν ούτε να... να... και θέλουν να αντισταθμίσουν απλώς τον λανθάνοντα επιχειρηματικό κίνδυνο. Θέλουμε ένα σταθερό σύστημα ε, που θα δίνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρειάζονται από την πραγματική οικονομία και θέλουμε να μας καθησυχάσετε ότι αυτές οι δραστηριότητες υπέρ του φόρου δεν θα δημιουργήσουν ένα συστημικό κίνδυνο και δεύτερον ότι θα βοηθήσουν για να, βοηθήσουν, να χτίσουμε πιο βαθιές και πιο ρευστέ αγορέ. Ξέρω ότι η συζήτηση του προτινόμενου φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, και το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ, συνδέεται με ένα μεγάλο αριθμό πολύ ευαίσθητων θεμάτων που συμπεριλαμβάνουν την επίπτωση στα χρηματοπιστωτικά κέντρα από την εφαρμογή του φόρου, την αποτελεσματικό του φόρου ε, στην εξασφάλιση κάποιας δημοσιονομικής αντιστάθμισης για το κόστος της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης και τη χρήση του φόρου για να αποθαρρύνουν δραστηριότητες που δεν έχουν προσθέμενη αξία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η οργάνωσή μας, η AECT που εκπροσωπώ, δεν θα εμπλακεί σε πολιτικές συζητήσεις ούτε ακόμα και αν υιοθετηθεί γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο φόρο, από όλε τι χώρε δηλαδή, ο φόρο αυτών των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Παρότι οι παρατηρήσει που θα ακούσατε μπορεί να σα κάνουν να πιστέψετε ότι εγώ προσωπικά αμφιβάλλω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει σύντομα. Οι βασικέ αρχέ που διαμορφώνουν τι απόψει των χρηστών του χρηματοπιστωτικού συστήματο, όπω εκπροσωπούνται από τα μέλη τη EACT, είναι οι εξή. Ότι καταρχά υποστηρίζουμε δράση για την ενίσχυση των κανόνων στο χρηματοπιστωτικό τομέα Δεύτερον, ότι ελπίζουμε ότι η συζήτηση για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα εστιάσει στο αν το κόστο του φόρου θα βαρύνει τελικά εσωτερικά το χρηματοπιστωτικό τομέα ή αν θα περάσει, θα μετακυληθεί πραγματικά στην ε, πραγματική οικονομία, τι εταιρείε, τα άτομα και στα συνταξιδοτικά ταμεία. Τρίτον, ελπίζουμε ότι θα μα καθησυχάσετε ότι οποιαδήποτε ανεπιθύμητη συνέπεια από την εφαρμογή του φόρου δεν θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση της αποτελεσματικότητας του νέου χρηματοπιστωτικού κανονιστικού περιβάλλοντος. Μετά από αυτές τις αρχές θέλω να τονίσω τρεις τομείς για συζήτηση γύρω από το, την πρόταση που αφορά το φόρο. Καταρχάς, ο σωρευτικός χαρακτήρας του φόρου μέσα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα δεδομένα από την BIS δείχνουν ότι τελικοί χρήστες ε, διενεργούν το ένα, ένα μικρό ποσοστό των συναλλαγών παραγόγων. Και με βάση εκτιμήσει, αυτό το ποσοστό είναι περίπου γύρω στο 5% και όχι στο 10%. Και τα νούμερα μάλιστα είναι σε... μειώνονται. Ε, μέσα στο σύστημα, πολλέ συναλλαγέ λαμβάνουν χώρα πριν ο τελικό χρήστη εμπλακεί. Ο προτινόμενο συντελεστή φόρου μπορεί να σα φανεί πολύ χαμηλό, αλλά η συσσόρευση του φόρου ε, μέσα στι τράπεζε τελικά οδηγούν σε ένα νούμερο πολύ ψηλότερο. Δεύτερον, σημείο προ συζήτηση. Εάν οι τελικοί χρήστε τελικά θα, βαρύ, θα φέρουν το, το βάρος, ε, το σωρευτικό βάρος του φόρου. Ε, διάφοροι σχολιαστές ε, συμφώνησαν ότι οι πελάτες των τραπεζών τελικά θα αντιμετωπίσουν υψηλότερο κόστος, καθώς οι τράπεζες θα προσπαθήσουν να κρατήσουν το περιθώριο κέρδους τους και να ανακτήσουν το, το φόρο αυτό. Και από την εμπειρία που έχουμε οι ταμείες εμείς από τις τράπεζες είναι ότι αν οι τράπεζες έχουν μια στεναρή στάση απέναντι στους πελάτες τους, ακόμη και πιο ισχυρές επιχειρήσεις δεν μπορέσουν να αντισταθούν. Τρίτο σημείο προ συζήτηση. Πώ θα αντιδράσουν οι τελικοί χρήστε. Η σημασία των παραγόγων για την αντιστάθμιση του κινδύνου από την πραγματική οικονομία είναι ότι χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν το τον λανθάνοντα κίνδυνο στη κλασική εμπορική δραστηριότητα και για τη χρηματοδότηση των τραπεζών. Μπορεί ε, οι τελικοί χρήστε λοιπόν να αντιδράσουν στο υψηλότερο κόστο με δύο τρόπου. Μειώνοντα τη χρήση των παραγόγων και αναδιοργανώντα τι δραστηριότητέ του, ούτω ώστε η αντιστάμιση του κινδύνου να συνεχιστεί χωρί να φέρουν οι εταιρείε του το άμεσο και άμεσο φόρο, ε, κόστο του φόρου. Και αυτέ οι δύο συνέπειε ήταν κακέ για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μείωση ε, του hedging, τη αντιστάθμιση του κινδύνου, ε, σημαίνει μεγαλύτερο κίνδυνο για την πραγματική οικονομία. Ε, Υψηλότερο κίνδυνο σημαίνει μεγαλύτερη προσοχή σε επενδύσει και σε επενδυτικέ αποφάσει, λιγότερα κέντρα για ανάπτυξη και απασχόληση. Η μετακίνηση των συναλλαγών επιπαραγόγων εντός, εκτός του, του πεδίου του φόρου αποδυναμώνει το ρυθμιστικό πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποσκάφει την πρόοδο που έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα. Πιστεύουμε ότι η πραγματική οικονομία πρέπει να προστατευθεί από τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις και οι τελικοί χρήστες, οι εταιρείε, τα άτομα, τα ασφαλιστικά και συνταξιωτικά ταμεία ε, δεν θα πρέπει να τους ζητήσουμε να φέρουν το βάρος από την επιβολή του φόρου. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε την Επιτροπή Σαστινιακών να ζητήσει μια εξαίρεση για τον τελικό χρήση από την εφαρμογή του φόρου και στις πραγματικές συναλλαγές και σε ό,τι αφορά την συσσόρευση του φόρου που συνδέεται με τις ε, δραστηριότητες του τραπεζικού τομέα πριν από την συναλλαγή με τους τελικούς χρήστες. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν τεράστιες πρακτικές ε, δυσκολίες ε, με αυτή την πρόταση. Πιστεύουμε όμως ότι με το να θέσουμε αυτή την αρχή μπορούμε να ενισχύσουμε ε, τη συζήτηση για, για να δούμε τελικά πού θα πέσει το βάρος από την εφαρμογή του φόρου αυτού. Σας ευχαριστώ και περιμένω να απαντήσω ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε και που τηρήσετε το χρόνο σας. Η κυρία Ποδηματά θα μιλήσει στο τέλος η συγκεκριά μας. Θα δώσω τώρα το λόγο στους και ηγητές. Εκ μέρους του ΕΛΚ θα μιλήσει πρώτα ο κύριος Φέρμπερ. Äh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακόμα τους επιγνώμονε, είχα την εντύπωση ότι ο φόρος χρηματοπικών συναλλαγών είναι το μαγικό φίλτρο που θα λύσει όλα τα προβλήματα που έχουμε μέχρι στιγμής αντιμετωπίσει. Και ακούγοντας κάτι τέτοιο βέβαια μου δημιουργούνται αμφιβολίες. Πρέπει να έχουμε κάποια θέματα κατά νου για να μην ε, βλέπουμε να διαπράττονται κάθε πράγμα, κάποια πράγματα αλλού και όχι εδώ και να εισαγάγουμε μόνο τα προβλήματα που απορρέουν από αυτές τις συναλλαγές. Είδαμε και στο παρελθόν θέματα που απήχαν πάρα πολύ από την ευρωπαϊκή οικονομία ξαφνικά είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και από τότε προσπαθούμε να διορθώσουμε. Έχουμε μη ομοιογενή χώρο νομισματικό, οικονομικό και κοινωνικό που προσπαθούμε να τους συνενώσουμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πετύχουμε αυτό που είχαμε καταρχήν κατά νου. Και τώρα προσπαθούμε το ίδιο να κάνουμε ένα κοινό φόρο. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Αν ήταν τόσο εύκολα θα το είχαμε κάνει εδώ και καιρό. Και γι' αυτό δεν μπορώ παρά να τονίσω κάτι που είδα σαν κύρια γραμμή όλων των ε, ομιλιών. Να δούμε καταρχήν τι κάνουμε. Καταρχήν, ποιον θα αφορά ο φόρος αυτός. Είναι πολύ απλό να αλλάξουμε το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, γιατί όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Αλλά δεν είναι αυτός ο τομέας ε, που χρειάζεται περισσότερο διακονισμό. γιατί έτσι ίσως φορολογούμε κάτι που δεν θέλαμε να φορολογήσουμε, όπως παραδείγματος χάρη συντάξει συντάξεις ε, και λοιπά. Είναι πολύ εύκολο βέβαια να φορολογήσουμε εκεί. Αλλά θα πρέπει να δράσουμε σωστά. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Παρόλο που θεωρώ ότι ο όρος φόρος στα γερμανικά τουλάχιστον, προέρχεται από την δυνατότητα κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη μας αυτό, ότι κάτι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό το φόρο. Κάτι θέλουμε να κάνουμε. Αλλά από την άλλη μεριά δεν θέλουμε μέσω φορολογικής νομοθεσίας, δηλαδή την φόρο για τις χρηματοπιστικές συναλλαγές παραδείγματος να διακανονίσουμε τόσο πολύ που να μην γίνεται πια τίποτα και όλες οι συναλλαγές αυτές να γίνονται κάπου αλλού πολύ πιο έντονα που δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο στόχος μας. Τρίτο πρόβλημα που θα ήθελα να έχουμε κατά νου και θα ήθελα να πάρω κάποιες απαντήσεις στο τέλος. Έχω την εντύπωση αυτή τη στιγμή ότι κάνουμε αυτό που κάνει παραδοσιακά η πολιτική όταν έχει ένα πρόβλημα εδώ και εμεί το κάνουμε διπλά στην Ευρώπη. Δηλαδή μια φορά σε ευρωπαϊκό και μια φορά σε εθνικό επίπεδο αναπτύσσουμε κάποιους κανόνες του παιχνιδού, διακανονισμού, εποπτείας και τώρα φορολογικές δυνατότητες. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή, να μην διακανονίσουμε τόσο πολύ, ούτως ώστε κάποια πράγματα που θα έπρεπε να λαμβάνουν χώρα, δεν λαμβάνουν χώρα. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί κυρίες και κύριοι και με την επικάλυψη εθνικών και ευρωπαϊκών διακανονισμών και ε, επιβολής φόρων που η κυριαρχία υπάρχει στα κράτη-μέλη, να μην πετάει λέω το αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο που επιθυμούμε. Και τέλος, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί φορολογικά έσοδα που δεν έχουμε ακόμα να μην τα δαπανούν ήδη. Δηλαδή άκουσα πολλά για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε το φόρο των χρηματοστών συναλλαγών. Λέω μπράβο, τόσα πολλά μπορούμε να εισπράξουμε και τι θα τα κάνουμε, τα ξέρουμε όλα. Και αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, εγώ λέω ξεκάθαρα, η κίνδυνη. Μία τελευταία πρόταση, κύριε Γιουσέρα τα κράτη-μέλη έχουν ε, το κύριο βάρος από την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και γι' αυτό θα πρέπει να είναι εκείνοι που θα αφαιρεθούν και περισσότερο. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Γιατί αν στο τέλο έχουμε την επιτυχία ενός τέτοιου φόρου θα ήταν πολύ καλό και κάτι που το επιθυμώ και εγώ ίδιος. Ευχαριστούμε κύριε Φέρμπερ. Θα σας διαβάσω το κατάλογο των ομιλητών. Γκίγκολ, Clute, señor Madeline, señora Hübner. Con esto... Ah. Shadows before. Shadows before. We'll speak before. But this is the... Πρώτα οι σκιώδεις. Προηγούνται οι σκιώδεις εισηγητές στη συζήτηση. One who may... Continuamos con el siguiente ponente en la... Επόμενος και ο είναι ο κύριο Κλίντ εκ μέρου των Φιλελευθέρων. Αλλά σα θέρμο παρακαλώ να περιοριστείτε σε δύο λεπτά γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μόνο δύο λεπτά καθ' ναι, ναι, ναι, ναι, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Μετά την ε, πτώση της Lehman Brothers, μέσα στα πλαίσια στο G20, αποφασίσαμε ε, κάθε ε, προϊόν, κάθε συμμετέχοντα συναλλαγές να την δεκανονίζουμε και ελέγχουμε και, χρηματο... και φορολογούμε τον ίδιο τρόπο. Ξέρουμε μετά από τέσσερα χρόνια ότι ακόμα απέχουμε πάρα πολύ. Υπάρχουν τεράστιε διαφορέ σε σημαντικού τομέα μεταξύ των ΗΠΑ και τη Ευρωπαϊκή και οπωσδήποτε άμα πάρω και την G20 μπορώ να συγκρίνω και με άλλες χώρες όπου οι διαφορές είναι ακόμη μεγαλύτερες. Γι' αυτό πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ούτως ώστε τουλάχιστον μέσα στους εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε μια ενιαία προσέγγιση, ιδίως όσον αφορά τους φόρους, ότι εδώ ήδη υπάρχουν διαφορές. Και στα πλαίσια αποφάσεων που λήφθησαν τελευταία έχουμε ένα φόρο στις τράπεζες, σε διάφορε χώρε που διαφέρει από χώρα σε χώρα ή και σε άλλε χώρε δεν υπάρχει καθόλου. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι εκ των προτέρων κατά του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αλλά θα ήθελα να πρωτοποιήσω μην εφαρμόσουμε το φόρο αυτό, εάν δεν είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε ενιαία ε, φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τουλάχιστον στον χώρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν τελικά ε, όπως είπε ο πρόεδρος Σαρκοζή τελικά το είπε θα το κάνω και μόνος μου και υπάρχει μόνο σε τρεις-τέσσερις χώρες τότε θα υπάρχει σαν αποτέλεσμα μια στρέβλωση και όχι ε, ενίσχυση της τουρκικής αγοράς που είναι ο κατά βάση στόχος μας και γι' αυτό θα έλεγα σαν στόχο να μην το παραβλέψετε αυτό. Ο τελευταίος ομιλητής εξέφερε τις αμφιβολίες του κατά πόσον αυτός ο φόρος, εάν εισαχθεί στην Ευρώπη, θα μπορέσει πραγματικά να εισαχθεί και παγκόσμια. Εγώ θα έλεγα αν συμφωνήσουμε οι 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τολμούσα να κάνω τη δοκιμή, ελπίζοντα ότι και άλλε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να μα ακολουθήσουν. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον τελευταίο ομιλητή. Θεωρεί ότι εάν η Ευρώπη ενωμένη εισαγάγει ένα τέτοιο φόρο, θα είναι αυτό ένα θετικό μήνυμα για το υπόλοιπο του κόσμου ή οι επιφυλάξει είναι μεγαλύτερε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καμάλ, εκ μέρου των συντηρητικών μεταρρυθμιστών. Σα ευχαριστώ. Ακούσαμε τα εισαγωγικά σχόλια όλων και ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε γιατί ε, ο φόρος ε, που είχε καταρχήν ε, προταθεί για τις ε, ενιαίες αγορές. Ε, ο Τόμπιν μπορεί να είναι μεγαλοφύη, αλλά ο φόρος Τόμπιν είναι πολύ ανόητος φόρος. Γιατί αν δούμε τα οικονομικά στοιχεία τι μας δίνουν, ότι πολλοί που κινδύνευαν από πτώχευση κάπως τακτοποιήθηκαν, καμία χώρα δεν απέφυγε την κρίση. Βρισκόμαστε γενικά σε μια κρίση. Έχουμε όλες αυτές τις προτάσεις, αλλά σήμερα, τρία χρόνια μετά την οικονομική κρίση, εάν μια τράπεζα φτωχεύσει μεθαύριο, θα ζητήσει χρήματα του φορολογούμενου για να ε, ορθοποδήσει εκ νέου. Δεν έχουμε λύσει αυτό το ουσιαστικό πρόβλημα, να είμαστε σίγουροι ότι αν μια τράπεζα πτωχεύσει να μην ζητάει χρήματα από τους φορολογούμενους. Λοιπόν, αυτό που ζητάω από ένα φόρο πιστικών συνολογών είναι κατά πόσο είναι θέμα που αφορά τις τράπεζες. Έχει επιπτώσεις στις τράπεζες. Ορισμένοι ψωμιλητές είπαν όχι. Ε, το κόστος μεταβάζεται στους ε, αποταμιευτές, ε, στις, ε, ε οργανισμούς κλπ. Τι θα γίνει λοιπόν. Πώς μπορεί κανένας να αποφύγει ε, ανεύθυνη συμπεριφορά των τραπεζών. Δηλαδή γιατί ε, πετάμε τα χρήματά μας σε χώρες που δεν μπορούν να συμβιβαστούν. Τι μήνυμα θα αποστείλουμε στους ε, πολίτες της Ευρώπης και αν τα χρήματα αυτά δοθούν σε αναπτυσσόμενε χώρε, πολλοί νομίζω θα χαιρόντουσαν για κάτι τέτοιο. Αλλά το θέμα είναι πώ μπορεί κανένα να αποφύγει να πάνε σε χώρε που έχουν κακή διαχείριση και τα χρήματα αυτά επανέλθουν σε ελβετικέ τράπεζε. Εάν θέλει κανένα να δει ποια είναι τα διδάγματα από την τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση, δεν θα έπρεπε να κάνει κάτι πιο ουσιαστικότερο. Να δούμε δηλαδή ποια είναι η ερμηνεία των προτύπων RFR που αγνοεί κάποιες αρχές δεν θα πρέπει να φροντίσουμε να αποκλείσουμε οποιαδήποτε ενίσχυση τραπεζών που βρίσκονται σε κατάσταση τόσο αυτής. Ναι, ναι, τελειώνω. Και να είμαστε σίγουροι οι διευθυντές των τραπεζών αυτών να είναι ε, υπεύθυνοι. Λοιπόν, ας ωφεληθούν από τις πλημμοδοτήσεις τους όταν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά θα αναλαμβάνουν την ευθύνη όταν πάνε καλά. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Πρασίνων, κύριο Καλφά. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβουμε τώρα τη συζήτηση περί κατά του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θα ήθελα να επανέλθω στα σχόλια των Φέρμπερ και κλιντ ε, Είπαν ότι θα υποστηρίξουν το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αρκεί να είναι παγκοσμιο Ναι, αλλά στη Γερμανία παρόλο που ήταν η μόνη που το εφάρμοσε, το ΣΥΔΕ ήταν κατά. Αυτό δεν εμπόδισε του άλλου έξι να το εφαρμόσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριο Κλίντ και το κόμμα του ε, συμμετέχει σε μια κυβέρνηση που μονομερώς με την Ελβετία ε, ενέκρινε τους φόρους Ρούμπικ. Ε, πολλά γίνονται δηλαδή και εντός των χωρών μελών που γίνονται στο εσωτερικό τους και όχι σε επίπεδο 27 πανευρωπαϊκά και παρόλα αυτά ε, τα υποστηρίξατε. Και τώρα για το φόρο χρηματοπιστώτησης συναλλαγών ξαφνικά και να είναι σε επίπεδο 27 αν είναι πανευρωπαϊκός. Τώρα, είναι μάλλον απίθανο η Βρετανική κυβέρνηση, εκτό και μα διαβεβαίωσε για το αντίθετο κ. Καμάλ, να δεχτεί έχει πρόθεσμα το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Το θέμα είναι, μπορούμε παρόλα αυτά να τον εφαρμόσουμε τουλάχιστον στην Ευρωζώνη. Και η ερώτησή μου προ του ε, προσκεκλημένου μα είναι τι αλλάζει στην θέσπιση του δικαίου και στην διατύπωση της οδηγίας αν αντί για εφαρμογή σε 27 χώρες ε, τον εφαρμόσουμε σε πιο στενό κύκλο, στην Ευρωζώνη ή και στις υπόλοιπε που θέλουν εκτός Ευρωζώνης. Ε, μια και βρισκόμαστε σε ενιαία αγορά. Έχουμε μια ενιαία αγορά 27 χωρών μελών και μια πρωτοβουλία που μπορεί να ληφθεί πιο περιορισμένα. Πώς θα λύσουμε αυτή, αυτές τις ε, εντάσεις. Και σε ό,τι αφορά την πρόταση των προσκεκλημένων να υπάρχει υποχρέωση για τις ε, μεταβιβάσεις τίτλων ε, ιδιοκτησίας, κυριότητας. Νομίζω ότι έτσι θα αποφύγουμε σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο μετακατάσταση. Ποια είναι η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γι' αυτό. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της ΓΚΟΕ τώρα, ο κύριος Πόρτας είναι ο σκιώδης ηγητής, αλλά απουσιάζει βλέπω. Δεν ξέρω αν κάποιος θα τον αναπληρώσει. Ο κύριος Κλούτε, Κλούτε συγγνώμη, για δύο λεπτά. Ναι, ευχαριστώ. Είχα ζητήσει το λόγο έτσι κι γιατί ε, τώρα μου το δείτε πιο νωρί. Είχα κάνει δύο παρατηρήσεις για τους τελευταίους ε, μελητέ του κ. Ρέμπορν που είπε ότι ο φόρος των προσωπικών συλλογών είναι κίνδυνο για την πραγματική οικονομία. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί για την πραγματική οικονομία ο πραγματικός κίνδυνος είναι η κρίση που αντιμετωπίζουν. Δηλαδή είχαν δυσκολίε να πάρουν δάνεια ο φόρος χρηματοσυμπιστικών συναλλαγών πρόκειται να σταθεροποιήσει τι αγορέ και να αποτρέψει αυτού του τύπου τη κρίση. Ε, δεν καταλαβαίνω λοιπόν το επιχείρημα, γιατί μακροπρόθεσμα θέλουμε να έχουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο η πραγματική οικονομία να μπορεί σωστά να αναπτυχθεί και να μην πλήττεται από αυτέ τι οικονομικέ κρίσει που ζήσαμε και ζούμε. Προ τον Μάρκο Φέρμπε. Είναι μόνο αναπληρωτή, αλλά είμαι στην Επιτροπή Προπολογισμών εδώ στο Σώμα. Και από ό,τι άκουσα, ο φόρο των προσωπικών συναλλαγών θα είναι έμεσα προ όφελο των κρατών μελών γιατί θα αυξήσει του ίδιου πόρου, Οι ίδιοι πόροι όμως θα συμβάλλουν ούτω ώστε οι άμεσε πληρωμέ των κρατών μελών θα μειωθούν. Αυτή τη στιγμή είναι σχετικά ψηλέ. Έμεσα λοιπόν θα είναι προ όφελο των κρατών μελών από ό,τι κατάλαβα στην Επιτροπή Προεπολογισμών. Θα συζητηθεί το θέμα αυτό, γιατί δεν κατάλαβα το επιχείρημά σα. Δύο ερωτήσει τώρα Καταρχήν, η ε, ε πρόταση κομισιόν εξαιρεί τις ε, συναλλαγές ε, λόγω της ελεύθερης κυκλοφορίας. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Υπάρχει στο Βέλγιο ένας νομικός που είπε ότι είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο να επιβάλλεται ο φόρος χρηματοστών συναλλαγών και στις ε, ε, συναλλαγματικές συναλλαγές. Δεύτερη ερώτηση. Εξέτασα το θέμα με συναδέλφους στην Γερμανία από το δικό μου κόμμα και μου είπαν ότι η υποχρέωση καταβολή φόρου μπορεί να αποφευχθεί εάν κανένα συνενώσει όλες τις αλλαγέ, και αύριο ε, τις κάνει εκτός του χώρου ε, ευρωζώνης εάν καταρχήσει εισαχθεί ο φόρος αυτός μόνο στην Ευρωζώνη. Αιματοποιεί, κάνει την αλλαγή του εκτός ε, Ευρωζώνης και μετά ξαναφέρνει τα κεφάλαια πίσω. Δεν ξέρω, είναι σωστό αυτό, δεν είναι σωστό. Τι πιστεύετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κλούτε. Τέλος, η κυρία Αντρίσεν έχει το λόγο για δύο λεπτά, η τελευταία σκιώδηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ με αυτούς που μιλήσανε προηγουμένω ότι το κύριο ουσιαστικό πρόβλημα που έχω με τον φόρο αυτό χρηματοστοπικών συναλλαγών είναι ότι η Κομισιόν τον πρότεινε το φόρο αυτό για να χρηματοδοτήσει τον ε, προπολογισμό της Ένωσης. Ε, αυτό που προσπαθεί να αποφύγει η Κομισιόν είναι οι διαπραγματεύσει που γίνονται κάθε χρόνο με τους αρχηγούς κυβερνήσεων των κρατών μελών για τον προπολογισμό της Ένωσης. Και αυτός ο φόρος που προτείνεται τώρα είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης του κοινοτικού προπολογισμού χωρίς προσπάθεια από τα κράτη-μέλη. Αλλά δεν είναι αληθές αυτό. Ή υπάρχει επικάλυψη. Δηλαδή οι φόροι που πληρώνουν αυτή τη στιγμή οι πολίτες των κρατών μελών θα παραμείνουν στα χέρια των κυβερνήσεων και εκτός αυτού οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να πληρώσουν ένα συμπληρωματικό φόρο για να χρηματοδοτήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαράδεκτο μου φαίνεται αυτό. Δεν μπορεί να αιτιολογηθεί κάτι τέτοιο. Δεν θα υπάρχει δηλαδή πια κανένα λόγο ή κανένα δυνατότητα εποπτεία και εξέταση στον λογαριασμό τη Ένωση, γιατί η κανενα δυνατοτητα εποπτεια και εξεταση των λογαριασμο Ένωση θα χρηματοδοτείται από το φόρο αυτό χωρί όρια ό,τι χρήματα θα παίρνουν θα τα χρησιμοποιούν. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που έχω. Γιατί δεν έχω ικανοποιηθεί ότι αυτό δεν θα επιβαρύνει τον, τελευταίο, τον τελικό χρήση. Ούτε έχω ικανοποιηθεί για το, όσα λέγονται για τον τρόπο με τον οποίο θα κατανοηθεί. Λοιπόν, ε, είμαι αντίθετη και νομίζω ότι ευθυγραμμίζομαι τον τελευταίο μιλητή.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 Merci beaucoup. Ahora damos la palabra a la Comisión Europea durante dos minutos. Por Si j'appuie, me regardez, normalement il y a un, plan. Oui, il y a Ça c'est quand Yeah, thank you very much, Mr. Chairman. Only a brief reaction to some of the speakers. Broad, more or less broad support the Commission proposal has got at this hearing.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 C'est bon Ένα, δύο. Ναι. Μεταξύ των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων. Σε ό,τι αφορά το risk hatching, δεν σημαίνει μείωση του κινδύνου. Θα πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν η αμερικανική κρίση ε, του subprime μετατράπηκε σε παγκόσμια κρίση. Ακριβώς ε, εξαιτία ε, του υψηλού κινδύνου ορισμένων προϊόντων. Μερικοί θεωρούσαν ε, ότι αγοράζοντα τα προϊόντα θα είχαν στα χέρια του προιοντα τριών 3α. Θα πρέπει κάτι που δεν ίσχυε στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να προσέξουμε όλα αυτά. Δεν πιστεύουμε ότι τα swaps μπορούν εύκολα να αξιολογηθούν με το δέλτα ή με άλλη μέθοδο. Θα πρέπει να βρεθεί και εκεί η σωστή μέθοδος για να αξιολογηθεί έκθεση κινδύνου στον κίνδυνο ενό προϊόντο. Δεν περιμένουμε από τι φορολογικέ αρχέ να επιστρέψουν χρήματα σε περίπτωση που αλλάξει το επίπεδο του κινδύνου. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι 80 με 90% ε, των, ε, των συναλλαγών είναι συναλλαγές μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Είναι δικοί τους δηλαδή οι πελάτες. Και όταν ε, βλέπουμε προϊόντα που είναι και τα πιο αποδοτικά είναι τα SOAPs και τα επιτόκια. Μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είδε καμία μελέτη που να δείχνει τα μακροοικονομικά ωφέλη του mushrooming, ε, του πολλαπλασιασμού, της έγκριξης τέτοιου είδους ε, συναλλαγών, δηλαδή τα swaps και τα επιτόκια. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή έχουμε επίγνωση ε, του γεγονότος ότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να υποβάλουμε μια τέτοια πρόταση, ε, να υποβάλλετε προτάσεις για να ενισχύσουμε τα, την προσέγγιση των τριών α για όλα τα προϊόντα, όλες τις αγορές και όλους τους φορείς. Και επίσης να δούμε πώς θα μειώσουμε τον κίνδυνο μετεγκατάστασης χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Όταν υπέβαλε ε, η Επιτροπή την πολιτική για το κλίμα του κλίματος, δεν ήθελε διαρροή ε, του άνθρακα και στην περίπτωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε διαρροή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κύριε Μπέργμαν. Το λόγο και τώρα ο εισηγητής τη ΟΚΕ, ο κύριος Πανιέρη. Παρακαλώ ένα λεπτό μόνο κύριε Πανιέρη. Είναι ο εισηγητής τη Οικονομική και κοινωνική Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην δική μας Επιτροπή ετοιμάζουμε μία γνωμοδότηση και εγώ είμαι εισηγητή αυτή τη γνωμοδότηση και στην Ολομέλεια της 29ης Μαρτίου θα παρουσιαστεί η έκθεση αυτή. Ελπίζουμε να χρησιμεύσει στις δικές σας εργασίες και στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήδη είχαμε κάνει, είχαμε ετοιμάσει δύο εκθέσεις, δύο γνωμοδοτήσεις τα περασμένα χρόνια, όπου είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την εισαγωγή ενός φόρου. Αυτή τη φορά βρήκαμε κάποια στοιχεία τα οποία βρίσκουμε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Η πρόταση της Κομισιόν εντάσσεται στο εσωτερικό ενός νέου συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποτίθεται ότι εξασφαλίζει αυτή την οικονομική ανεξαρτηρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπει το 201 της συνθήκης της, προέβλεπε μάλλον το 201 της Ρώμης. Ένα νέο σύστημα λοιπόν που προβλέπει για την ε, με την εισαγωγή του φόρου 57 δις θα προέκυπταν, όπου τα 35 ε, θα πήγαιναν, 37 συγγνώμη, θα πήγαιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπόλοιπα 20 στα κράτη-μέλη. Ο φόρος αυτός ε, εισάγει μία τροποποίηση στον τρόπο λειτουργίας των εμπορευομένων και πλήττει τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας, που είναι πάρα πολύ κερδοσκοπικές και που δημιουργούν ε, αστάθεια στις αγορές. Μην ξεχνάτε ότι αυτό το μέσο μαζί με την καλύτερη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματαγορών θα επέτρεπε σε αυτούς τους τελευταίους, σε τις αγορές δηλαδή, να παίξουν να παίξουν το ρόλο τους και να βοηθήσουν και την πραγματική οικονομία. Παρακαλώ, μπορείτε να τελειώσετε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι από το 2010 οι Ευρωπαίοι πολίτες που είπαν ότι είναι υπέρ της εισαγωγής ενός τέτοιου φόρου ποτέ δεν κατέβηκε κάτω από το 60% με βάση, τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου. 60% των Ευρωπαίων πολιτών είπαν ότι είναι υπέρ. Ευχαριστούμε κύριε Παλμιάρη. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στους προσκεκλημένους μας για δύο λεπτά στον καθένα. Και πρώτα στον κύριο Περσότ. Αλλά παρακαλώ πραγματικά τηρήστε ευλαβικά το δίλεπτο. Ευχαριστώ. Θα χρησιμοποιήσω το δίλεπτό μου για να οριοθετήσω κάπως τη συζήτηση. Ο φόρος χρηματοπιστωτικός συναλλαγών δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τη χρηματοπιστωτική ρύθμιση, τη ρύθμιση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί και η ρύθμιση αυτή, ώστε να περιοριστεί η κρίση που είχαμε μέχρι τώρα. Και αν αναθεωρήσουμε το Βασιλεία 2, ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών συνάδει με το Βασιλεία 2. Γιατί ε, ξέρεις κεφαλαίο από βρακυπρόθεσμες ε, ε, δραστηριότητες μετατέθονται και ενθαρρύνει μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών. Είναι η Βασιλεία 2 συνεπής με το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και πολλά από τα επιχειρήματα που ακούσαμε σήμερα θα μπορούσαν να είχαν ισχύσει και για το φόρο εισοδήματο ή τον εταιρικό φόρο ή τι κοινωνικέ εισφορέ. Λέμε πώς θα αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα, πόσο θα ενθαρρύνει μια σωστή νοτροπία η τον εταιρικο φορο η τι κοινωνικε εισφορε λεμε πω θα αυξηθουν τα φορολογικα εσοδα ποσο θα ενθαρρυνει μια σωστη νοοτροπια η φορολογια και θα εξοβελήσει την λιγότερη αποδοτική δραστηριότητα. Και νομίζουμε ότι ενθαρρύνουμε περισσότερο τις μακρο μακροπρόθεσμες επενδύσεις εις βάρος των βραχυπρόθεσμων. Και είμαστε και συνεπείς με τις παραδόσεις και την ιστορία της Ευρώπης. Η επιτυχία της Ευρώπης σε μεγάλο βαθμό στηρίχθηκε στην οικονομία γιατί επένδυσε στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις ε, από ότι στις βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες. Είπαν μερικοί να περιμένουμε να συμφωνήσει και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μα ήδη έχει συμφωνήσει. Έχει έναν ποσοστό, ένα φόρο σε εναλλαγό 0,5% και εξακολουθεί το Λονδίνο να είναι η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική αγορά για δραστηριότητε hedging κεφαλαίων κινδύνου και επίσης θέλουμε να κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου. Θα πρέπει να αποφύγουμε τη, τα φαινόμενα φοροδιαφυγής. 40% των φόρου στο Ηνωμένο Βασίλειο καταβάλλεται από ολοδαπούς που φοβούνται να, ότι θα χάσουν τους τίτλους κυριότητάς τους αν δεν καταβάλουν αυτό το φόρο το τέλος χαρτοσύμου. Το Λονδίνο, το Χονγκ Κονγκ και η Ζηρίχη εφαρμόζουν φόρους χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και παρόλα αυτά εξακολουθούν να παραμένουν ε, τα πιο ανθυρά χρηματοπιστωτικά κέντρα διεθνώς. Ευχαριστούμε κύριε Πέρσο. Ο κύριος Καπούρ για δύο λεπτά. Ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι το αντιστάθμισμα των ε, ρυθμίσεων που ίσχυσαν στον τραπεζικό τομέα. Αν δείτε τους τραπεζικούς φόρους που έχουν εφαρμοστεί στο τραπεζικό σύστημα, βλέπετε ότι ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι το φυσικό αντιστάθμισμα της ε, κατάστασης και τώρα όπως βλέπετε θα φτάσουμε σε ένα καλώς ρυθμισμένο σύστημα το επίσημο δηλαδή τραπεζικό σύστημα. Αλλά το σκιώδες τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Γι' αυτό ακριβώς ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι ένα καλό μέσο προς αυτή την κατεύθυνση. Και οι επιπτώσεις θα ισχύσουν στο σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Όχι στην πραγματική οικονομία, στο επίσημο τραπεζικό σύστημα δηλαδή. Η πρόταση της Επιτροπής μιλά για ένα ελάχιστο ποσοστό. Και το ίδιο ισχύει και με τον ΦΠΑ. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα. Υπάρχει η βάση, αλλά οι ποσοστιαίες αναλογίες διαφέρουν και ίσως κάποια στιγμή συγκλίνουν. Το MIFID 2 και το ΕΜΙ που απασχολεί εμάς τώρα αποτελεί τη βάση εφαρμογής ενός τέλους, ενός φόρου. Είτε πρόκειται για ευρωπαϊκό επίπεδο, για Ηνωμένο Βασίλειο, χρειάζεται η νομιμότητα την οποία έχουμε, πληροφορίες και πιστεύω ότι το MIFID 2 και το EMIT πληρούν αυτούς τους όρους. Επίσης, θα πρέπει να αρχίσουμε με τις αγορές ομολογιών, μάλλον αρχήν με τα χρηματιστήρια, με τοχές ομολογίες και ούτω καθεξής. Μπορεί κανείς να αρχίσει με χαμηλότερο ποσοστό, να προβεί σε μια μελέτη αντικτύπου και μετά να δει ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος. Ευχαριστούμε κύριε Καϊπούρ. Griffith Jones. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολλοί ευρωβουλευτές πολύ σωστά τόνισαν ότι χρειαζόμαστε στην Ευρώπη ε, ένα χρηματοπιστωτικό τομέα που να εξυπηρετεί την πραγματική οικονομία. Να μην είναι κακός, ε, κακό αφεντικό, αλλά καλός υπηρέτης. Και Αν δεν το πετύχουμε αυτό στην Ευρώπη, δεν θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε την Ινδία, την Κίνα, τη Βραζιλία, που έχουν αποτελεσματικούς χρηματοπιστωτικούς τομείς, λιγότερο περίπλακους, περισσότερο διαφανείς, καλύτερα ρυθμιζόμενους θα πρέπει αυτό το φόρο να το δούμε σε αυτό το πλαίσιο. Ο σκοπός μας είναι να μεταρρυθμίσουμε το χρηματοπιστωτικό τομέα και να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Μου έκανα μια ερώτηση. Ότι θα ήταν πολύ άσχημο να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο φόρο ε, για, και να βάλουμε τα λεφτά αυτή, αυτά στην πράσινη οικονομία. Δεν νομίζω. Καταρχά θα, θα ήταν καλό για την ε, ανάπτυξη και την απασχόληση, γιατί μία πράσινη τεχνολογία είναι το μέλλον. Αν επενδύουμε σε τέτοιε τεχνολογίες, όχι απλώς ε, θα βοηθήσουμε να σωθεί ο πλανήτη, αλλά θα συνεισφέρουμε σε μια νέα βιομηχανική επανάσταση που θα έρθει. Υπάρχουν φυσικά εξωτερικές παράμετροι και στοιχεία που θα πρέπει εν μέρη να επιδοτηθούν από δημόσιους πόρους. Αλλά μακροπρόθεσμα θα έχουμε ε, μεγάλα οικονομικά ωφέλη θα έχουμε καταρχάς ένα πλανήτη για τα εγγόνια μας και τα δυσεγγονά μας. Κάτα, κάτι άλλο για τις παρακάμψεις. Ε, εγώ ήμουν στην πρώτη συζήτηση με τον James Tobin ε, και είχε πει ότι όταν εισήχθη για πρώτη φορά ο φόρος εισοδήματος είχαν ακουστεί επιχειρήματα περί φόροδιαφυγής. Και φυσικά υπάρχουν φοροδιαφυγές, αλλά είναι ακόμα καλός φόρος. Μάλιστα, όπω λέμε στο εγγραφό μα στι ΗΠΑ, έχουμε φοροδιαφυγή ύψου 18%. Παρ' όλα αυτά, μαζεύουμε 500 δι ευρώ και είναι προοδευτικό φόρο. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να το σκεφτούμε ε, με έναν τρόπο τόσο ώστε να τον σχεδιάσουμε με σκοπό να μειώσουμε όσο μπορούμε στο ελάχιστο τι φοροδιαφυγέ. Μπορούμε να συγκεντρώσουμε πολλού πόρου, πολλά χρήματα και παράλληλα μπορούμε να το σχεδιάσουμε έτσι ούτως ώστε να μην επηρεάσουμε την, αρνητική, την ε, πραγματική οικονομία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ριμπέρν, πολύ σύντομα. Ε, λέτε ότι ο φόρος ε, χαρτοσύμου είναι φόρος ε, FTT, ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Όχι, δεν είναι σωστό, γιατί δεν ε, ε, φορολογεί τι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ στο τραπεζικό τομέα. Ε, με ρωτάτε, ε, αν είμαι υπέρ του φόρου αυτού. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι δυστυχώς θα εφαρμοστεί παγκόσμια. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ε, και τέλος, αυτό που ο κ. Λάμπερτς είπε, ότι εγώ είπα, ότι οι ρυθμίσεις δεν θα πρέπει να αγγίξουν την πραγματική οικονομία. Όχι, δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι η ρυθμίση του χρηματοπιστωτικού τομέα δεν θα πρέπει να έχει αθέλητες συνέπειες, ανεπιθύμητες συνέπειες στην πραγματική οικονομία. Αυτό λέμε, αυτό ε, θέλουμε να αποφύγουμε, αυτό είναι το επιχείρημά μας. Είπε ότι τα παράγωγα ε, τα επινοήσαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Όταν, κύριε Λάμπερτς, ήσασταν αγοράκι, εγώ χρησιμοποιούσα παράγωγα. τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε χρησιμοποιήσει για πάρα πολλά χρόνια. Τέλος, είπατε ότι είναι 0,01% συντελεστής. Είναι 0,02% καταρχά. Ε, γιατί πληρώνουν και τα δύο μέρη της τελικής συναλλαγής. Και επιπλέον αυξάνεται μέσα στο σύστημα, καθώς ας πούμε οι τράπεζες κάνουν τα κακά πράγματα που κάνουν συνήθως οι τράπεζες, ε, σεωρεύεται ο φόρος αυτός. Οι πελάτες πληρώνουν και η πραγματικότητα είναι ότι θα πληρώσει και η πραγματική οικονομία. Δεν ξέρω τι θέλουμε να επιτύχουμε. Ευχαριστούμε κύριε Ράμπερν. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Ποδηματά. Για... Παρακαλώ. Πέντε λεπτά κυρία Ποδηματά. Σας θέλω παρακαλώ αν μπορείτε να περιοριστείτε σε πέντε λεπτό. Ε, προσπαθήσω να περιοριστώ στο χρόνο των πέντε λεπτών. Ήθελα πρώτα απ' όλα να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω θερμά και εγώ από την πλευρά μου όλους τους ε, εμπειρογνώμενες που συμμετείχαν ε, σε αυτή τη δημόσια ακρόαση, όπως και τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Ήταν άλλη μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και παραγωγική συζήτηση σε σχέση με την εισαγωγή ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ε, δεδομένου του περιορισμού του χρόνου θα κατηγοριοποιήσω τα ζητήματα που τέθηκαν και από τους εμπειρογνώμονες και οι εισηγητές μας και από τους συναδέλφους και θα προσπαθήσω να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα και σε κάποια σχόλια βεβαίως από τη δική μου πλευρά. Πρώτα απ' όλα, ε, από πολλούς συναδέλφους και από τους συζητητέ μας τέθηκε το θέμα τι θέλουμε να πετύχουμε ε, προτείνοντας την εισαγωγή ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Τι επιδιώκουμε με αυτό το φόρο. Και ε, είναι προφανές, το είπε και ο κ. Φάμπερ, ότι ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν είναι μια μαγική λύση που θα λύσει όλα τα προβλήματα, ούτε είναι σωστό να αντιμετωπίζετε και να θεωρείτε ε, τέτοια. Ε, από την άλλη πλευρά όμως νομίζω ότι μπορεί κανείς να καταλήξει στο συμπέρασμα από τις παρεμβάσεις των περισσότερων επιρρογνωμόνων και ομιλητών ότι ένας φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που θα εφαρμόζεται στην ευρύτερη δυνατή κλίμακα και θα έχει έναν ε, χαμηλό συντελεστή μπορεί να διασφαλίσει σημαντικούς πόρους για τους εθνικούς προϋπολογισμούς, για τη μείωση των ελλημάτων που αντιμετωπίζουν η συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών πολιτικών στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, με δικαιότερο τρόπο όλα αυτά. Με δικαιότερο τρόπο τι θα πει, θα πει με τη συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα, δηλαδή ενός τομέα που έχει ευθύνη, κατά την αποκλειστική, κατά τη βασική, κατά απλώς κάποια ευθύνη. Αλλά αναμφισβήτητα ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει ευθύνη για τη σημερινή κρίση, απολαμβάνει παρόλα αυτά πολλών προνομίων, μεταξύ των οποίων την εξαίρεσή του σε μεγάλο βαθμό από τη φορολογία. Άρα λοιπόν ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών διασφαλίζει μια δίκαιη συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα στο κόστο τη κρίση τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών ε, πολιτικών, ώστε να μην επιβαρύνεται συνεχώ και συστηματικά η εργασία και η παραγωγική οικονομική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει δικαιότερη κατανομή των βαρών και θέλω να πω με την ευκαιρία ότι όσοι ανησυχούν ότι τελικώς θα επιβαρυνθούν οι τελικοί καταναλωτές, τα νοικοκυριά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επειδή ο φόρος θα μετακυλιστεί όπως λένε, νομίζω ότι είτε ότι δεν ανησυχούν ειλικρινά, είτε ότι διαστευλώνουν την πραγματικότητα. Δεύτερο σημείο, ποιους θα επιβαρύνει ο φόρος. Θα επιβαρυνθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, θα περιοριστεί η ρευστότητα μειώνοντας τις συναλλαγές παραγόγων αντιστάθμισης κινδύνου, όπως αποδεικνύει και η μελέτη που έχουν συντάξει οι υπερογνώμονέ μας. Ε, δεν θα επιβαρυνθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, διότι τα ασφαλιστικά ε, ταμεία, μιλώντας με αριθμούς και με στοιχεία, κάνουν μία επενδυτική συναλλαγή κατά μέσο όρο μία φορά κάθε δύο χρόνια και αλλάζουν ε, το μισό ε, χαρτοφυλάκιο που διαθέτουν. Ε, ενώ ένας έμπορος υψηλής συχνότητας, ένας high frequency trader που αλλάζει ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό του στη διάρκεια μιας μόνο μέρας, είναι προφανές ότι αυτό θα επιβαρυνθεί από το φόρο, θα πληρώσει χίλιε φορέ περισσότερο κατά αναλογία και κατά τη από ότι το ασφαλιστικό ταμείο. Και εν πάση περιπτώσει δεν θέλουμε ασφαλιστικά ταμεία που κάνουν επενδυτικές επιλογές υψηλού ρίσκου, διότι και ε, τους πόρους τα κεφάλαιά τους θέτουν σε κίνδυνο και συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση του συστημικού ε, κινδύνου. Τρίτο σημείο. Μπορεί μόνος του ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών να, ε, να δημιουργήσει μια καλύτερη, ε, καλύτερους κανόνες ρύθμισης και εποπτείας στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Προφανώς και όχι. Αλλά αν μπορούμε σήμερα, όπως είπε και η κυρία Στέφανη ε, Γκρίφιθ Griffith-Jones σήμερα είναι ακριβώς η στιγμή για να μιλάμε για την εισαγωγή ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ακριβώς διότι σήμερα έχουμε κάνει σημαντικά βήματα δεν έχουμε καταφέρει τα πάντα, αλλά έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για ένα καλύτερο και ισχυρότερο πλαίσιο ε, ρύθμισης και εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Σήμερα, για παράδειγμα, ε, μιλάμε για νέους κανόνες στην αγορά των έξω χρηματιστηριακών παραγόγων. Είναι μια ρύθμιση που δεν την είχαμε μέχρι πρότινος και που μας δίνει τη δυνατότητα σε συνδυασμό ε, με την πρόταση για την εισαγωγή ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών πραγματικά να επικεντρώσουμε σε αυτό που λένε και οι εμπειρογνώμονές μας, που είναι και ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής, δηλαδή να περιορίσουμε, να αποθαρρύνουμε, να δημιουργήσουμε αντικίνητρα για εκείνες τις συναλλαγές που δεν έχουν καμία προσθέμενη αξία για την πραγματική οικονομία, που δημιουργούν ή ενισχύουν, πολλαπλασιάζουν τον συστημικό ε, κίνδυνο και να συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο και μαζί με τα υπόλοιπα εργαλεία, όπως έλεγα και πριν, στην επαναφορά του χρηματοπιστωτικού τομέα στο βασικό του ρόλο που είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και φτάσαμε στο τέλος της ακροάσης μας. Ευχαριστούμε τους εμπειρογνώμονές μας και όλους τους ε, μιλητές που έλαβαν μέρος σε αυτή την πολύ έντονη συζήτηση. Μην ξεχνάτε τη διορία για τις τροπολογίες που λύγει στις 3 Μαρτίου. Και περνάμε στο επόμενο σημείο, την εξέταση των τροπολογιών της ετήσιας έκθεσης του, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η συγητής μας είναι ο κύριος Καμάλ. Κύριε Καμάλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι για την καρποφόρα συζήτηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τους κοιόδης συγητές και ελπίζω η γνωμοδότηση της ε, ΚΟΝ να στείλει τέτοια είδους μηνύματα, τέτοιου είδους μηνύματα σύμπνοιας. That's right. Παρακαλώ, εκενώστε την αίθουσα όσο πιο γρήγορα γίνεται για να συνεχίσουμε. Είναι παράδεκτο. Οι θεατές να συνεχίζουν εδώ τις ιδιωτικές συνομιλίες και να μην εγκαταλείπουν την αίθουσα τάχιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Λεγκοζές. Συνεχίστε, κύριε Καμάλ. Ευχαριστώ. Ε, εγώ ήμουν βέβαιος ότι όλοι θα περίμεναν διακαώς να ακούσουν την παρέμβασή μου και πραγματικά θα χάσουν πάρα πολλά που φεύγουν. Χαίρομαι για την καρποφόρα συζήτηση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα με τους σκιώδεις ηγητές και ελπίζω ότι θα είναι χειρό το μήνυμα της, ε, της γνωμοδότησής μας. Οι πολιτικές ομάδες είναι υπέρ της διαφάνειας και της λογοδοσίας και θα πρέπει οι ΕΤΕ και οι δραστηριότητε τη να ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική του 2020 και επίση ε, να συνεργάζεται με την ΕΤΑ, την BERT για να μην υπάρχει επικάλυψη ε, των ε, κονδυλίων. Θέλουμε βέβαια η ΕΤΕΠ να τηρήσει τα, τις προδιαγραφές της Βασιλείας 2 σε ό,τι αφορά την ε, επάρκεια κεφαλαίων και να είναι συνεπή, συν, ε, και με τη Βασιλεία 3. Θα πρέπει οι πολίτες να μπορούν να εντοπίζουν με ποιο τρόπο και πού δαπανώνται τα χρήματά τους και θα πρέπει αυτές οι πληροφορίες να δίνονται με διαφάνεια και να είναι προσιτές. Αυτός είναι ε, ο στόχος, το ζητούμενο για την ΕΤΕΠ. Οι σκιώδεις ηγητές είναι υπέρ της πρόθεσης των ευρωομολόγων προκειμένου να ενθαρρύνει τις ιδιωτικές ε, επενδύσεις στις ε, υποδομές. Επίσης υπήρχε υπερκομματική υποστήριξη του να ε, εστιάσει η ΕΤΕΠ τις δραστηριότητες στις χώρες της Βορειοαφρικής που βρίσκονται σε μεταβατική διαδικασία, σε διαδικασία εξυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού. Ευχαριστώ και πάλι τους και οδησηγητές για τις πολύ επικοδομητικές συζητήσεις που είχαμε και αν μου διέφυγε τίποτα από τη συνεδρίαση ελπίζω να το ακούσω τώρα για να το προσθέσουμε. Ευχαριστώ κύριε Καμάλ. Το λόγο έχουν τώρα οι σκιώδεις Ξεκινούμε από την κυρία Κράτσα από το ΕΛΚ. Δύο λεπτά παρακαλώ μόνο. Κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή διότι μας έδωσε ήδη με το προσχέδιο που υπέβαλε μια καλή βάση να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε την τελική μας ε, πρόταση. Ε, να τον ευχαριστήσω επίσης με το θετικό πνεύμα το οποίο αντιμετώπισε τις τροπολογίες μας. Ε, ανέφερε ήδη ο εισηγητής βασικές γραμμές που αποτελούν αποτέλεσμα των συμβαστικών προτάσεων που έχει υποβάλει και οι οποίες καλύπτουν και του ομάδα της ομάδας μας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Τροπολογίε και, και προτεραιότητες. Ε, επίσης θέλω, όπως η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ε, ε τη συνεργασία με τα διαφορετικά ταμεία ε, για να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τα εργαλεία μας και τα κέρδη μας ε, και επίσης τα, τα ομόλογα έργων, δέσμευση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, από την οποία περιμένουμε πολλά ε, ε, ε, τον έλεγχο της χρηματοπιστωτικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είναι βασικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στις δικές μας απόψεις. Επίσης θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί βλέπει θετικό πνεύμα ε, και άλλα θέματα τα οποία έχουμε υποβάλει εμεί ως ιδέες, παραδείγματο χάρη να διελευκανθεί η θέση της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων σε σχέση με το ΦΕΜΙΠ, το εργαλείο Ανάπτυξης ε, της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, το οποίο ήδη υπάρχει. Επίσης, τη σημασία στα προγράμματα Jessica, Jeremy, Jasmine, Jaspers είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη, την περιφερειακή και τη συνοχή επίσης, μια άλλη παρέμβαση που κάνουμε είναι η έμφαση και η ενθάρρυνση της καινοτομίας, ε, της έρευνας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και ε, ο εισηγητής το λαμβάνει υπόψη του. Και επίσης ε, η, η παρέμβαση στις χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές δυσκολίες είναι ήδη για την Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων μια πραγματικότητα και δίνουμε έμφαση και εμείς στο, στην, στις τροπολογίες μας πως μέσω των διαχρονικών ταμείων, της υποστήριξης στη χρηματοδότηση των διαφορετικών ταμείων θα ευνοήσει ε, η τράπεζα την ε, ε, έξοδο από την κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτά ήθελα να τονίσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κράτσα. Το λόγο κύριος για δύο λεπτά. Ε, ε, Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καμάλη για την πολύ καλή συνεργασία μέσω αυτής της έκθεσης. Θα ήθελα να πω ότι φτάσαμε σε συμβιβασμούς που είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι και ανάμεσα σε αυτές τις τροπολογίες θα ήθελα να αναφερθώ στην ενθάρρυνση του συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ ΕΤΕ και Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Επίσης, ε, συμβαδίζουμε με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τουλάχιστον προσπαθούμε μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας των ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου, επίσης πολέμηση των φορολογικών παραδείσων και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, πριν από την έγκριση ενός σχεδίου θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ελέγξουμε με διαφάνεια τις διάφορες περιφέρειες που θα ευεργετηθούν από τους πόρους αυτούς. Επίσης, να προσπαθήσουμε να προβάλλουμε μελέτες αντικτύπου και τέλος την εφαρμογή των σχεδίων, μάλλον την αναπρότζεκτ προσέγγιση και χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Χρειαζόμαστε η οικονομική ανάπτυξη, μόνιμη οικονομική ανάπτυξη και πιστεύω ότι θα πρέπει στα πλαίσια των διευρωπαϊκών δικτύων της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της έρευνας να δοθεί ένα κίνητρο έτσι ώστε να ε, προωθηθούν αυτά τα πρόγραμματα. Σας ευχαριστώ κύριε Κούτας και επειδή αρκεστήκατε στο χρόνο, η κυρία Γκουλάρ έχει το λόγο. Από τους φιλελεύθερους δύο λεπτά. Ο κύριος Χιλακάκης δεν είναι εδώ ε, τον αντικαθιστώ και θέλω να σας πω ότι η δουλειά ήταν πολύ επικοδομητική. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Δεν έχουμε ιδιαίτερε παρατηρήσει, ε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειε λοιπόν. Θέλω απλώ να τονίσω ότι για την ομάδα μα, όπω είπαμε και ξαναείπαμε και στην Ολομέλη ακόμα, ο Γκί το είπε μάλιστα, η ιδέα ότι η ΕΤΕ μπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις ε, για το μέλλον μέσω των project bonds, μέσω των ομολόγων έργου, είναι πάρα πολύ σημαντική ιδέα, την υποστηρίζουμε ολόθερμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Γκουλά. Από τους πράσινους, ο κύριος Γκίγκολτ για δύο λεπτά. Σύντομα, ε, αντικαθιστώ τον Πασκάλ. Ε, σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία. Υποστηρίζουμε τους συμβιβασμού όπως τους παρουσιάσατε. Υπάρχουν κάποια θέματα ίσονος σημασίας που θα θέλαμε να συζητήσουμε, αλλά δεν είναι πολιτικής φύσεως, είναι μάλλον τεχνικής φύσεως. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία ακόμα μια φορά. Τέλος. Από την ΚΟΕ ο κύριος Κλούτ. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν θα επαναλάβω λοιπόν όσα υπόθηκαν. Δεν έχω να προσθέσω και πολλά. Αρκούν αυτά. Α, τέλεια, ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ο εκπρόσωπός θα μιλήσει για δύο λεπτά. Μία μικρή παρατήρηση. Μην ξεχνάτε ότι θέλετε η ΕΤΕ να κάνει νέες επενδύσεις. Υπάρχει όμως το πρόβλημα της, του δυναμικού της ΕΤΕ και της ικανότητάς της. Ε, θα πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε το δυναμικό της. Ε, υπάρχει ο κίνδυνος γιατί η, μόνο το δυνητικό κεφάλαιο λήφθηκε υπόψη από τις εταιρείες βαθμολόγησης. Πρέπει να πάρουμε το πραγματικό κεφάλαιο. Βλέπουμε επίσης ότι τα κράτη-μέλη της ΕΤΕ δεν είναι ε, σε θέση σήμερα έτσι όπως έχουν τα οικονομικά τους να δώσουν ε, τα επιπλέον κονδύλια που χρειάζεται η ΕΤΕ. Δεν ξέρω αν ο εισηγητής σκοπεύει να πει κάτι από αυτού, αλλά χρήσιμο θα ήταν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε ο εκπρόσωπο τη ΕΤΕΠ, τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστώ τον κύριο Καμάλ για την εξαιρετική του έκθεση και τον ευχαριστώ και για την συνεργασία. Και φυσικά ευχαριστήσει και προς τους και ηγητές και όσους κατέθεσαν τροπολογίες. Συνεχίζοντας ε, ε, αυτά που είπαμε τελευταίως προαλήσατες, αυτή, ακριβώς αυτή την ισορροπία ζητάμε μεταξύ του ρόλου του ΕΤΕΠ να επεμβαίνει και να στηρίζει τις κινητικές πολιτικές στους τομείς που αναφέρθηκαν, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποδομές, ε, περιβάλλον, κλιματικές αλλαγές και φυσικά να διαφυλάξει τα τρία αλφα και να κρατήσει το επιχειρηματικό της μοντέλο. Και γι' αυτό θα πρέπει ε, να δούμε πώς αντλούμε τα κονδύλια από τις χρηματοπιστωτικές αγορές ε, και πού δανείζουμε φυσικά με όσο δυνατόν υψηλή βαθμολόγηση ώστε να έχουμε πρόσβαση τα μία, το θεσμικό, στα κονδύλια των θεσμικών επενδυτών που είναι περισσότεροι δανειστές μας και ε, να μπορέσουμε το οικονομικό πλεονέκτημα του τριπλού α να το μεταλαμπαδεύσουμε στις χώρες μέλη και στους ιδιώτες ε, πελάτες μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Και φυσικά ασκήθηκε πίεση από τους οίκου αξιολόγηση και ε, πίεση στα κράτη-μέλη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε τα τρία α Αυτό είναι σημαντικό για το επιχειρησιακό μας μοντέλο. Τώρα για τα υπόλοιπα σημεία Έχουμε στενή συνεργασία με την BERT, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και όλο και περισσότερο επεκτείνουμε ε, τις, δραστηριότητε τις δραστηριότητες μας στη Μεσόγειο που θα περιληφθεί στο μνημόνιο συνεννόηση που είχαμε συνάψει πέρσι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τα project bonds, αυτά τα ομόλογα δεν είναι ομόλογα της ΕΤΕΠ ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ομόλογα των, ε, που εκδίδονται από τις ίδιες επιχειρήσεις ε, ε, που εφαρμόζουν, που εφαρμόζουν αυτά τα σχέδια υποδομών. Εμείς χρηματοδοτούμε τα δάνεια με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται σε πειραματική φάση αυτό το σχέδιο σε ό,τι αφορά ε, τα χρηματοπιστωτικά κέντρα και τα, τις ε, δικαιοδοσίες που δεν είναι και πολύ συνεργάσιμες εφαρμόζουμε τα αυστηρά κριτήρια. Και τέλος θα ξαναδώσω το λόγο στον ε, εισηγητή μας, τον κύριο Καμέλ. Ευχαριστώ και να ευχαριστήσω και πάλι τους, συγητές, ε, τους για τα ευγενικά του σχόλια. Ε, δεν χορταίνω αυτά τα εγκόμια και τους επένους και την ευγνωμοσύνη. Συνεχίστε, συνεχίστε να με στολίζετε. Ελπίζω να συνεχίσουμε την επικοδομητική μας συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Καμάλ. Μην ξεχνάτε ότι θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή τη Δευτέρα, 13 του μηνός, 13 Φεβρουαρίου, στο Στρασβούργο. Και ερχόμαστε στο τελευταίο σημείο της ημερήσια διάταξη ε, εξέταση των τροπολογιών σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού. Η συγκεκριά μας είναι η κυρία Μπασέσκου και της δίνω το λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη γιατί είναι πολύ αργά. Όταν συναντηθήκαμε στις 19 Δεκεμβρίου υπέβαλα σχέδιο πρότασης για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Διαχείρισης Λογαριασμού. Πρόκειται για μια πολύ καλή πρωτοβουλία έτσι ώστε οι πιστωτές να μπορέσουν να ανακτήσουν τα χρήματα σε οποιοδήποτε λογαριασμό που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 27 τροπολογίες αφορούν σημεία διευκρίνηση του σχεδίου κανονισμού έτσι ώστε ε, να προβώ σε μία εξορρόπηση μεταξύ δικαιωμάτων ε, πιστωτή και οφειλέτη. Και άλλοι συνάδελφοι υπέβαλαν τροπολογίες, 11 τροπολογίες ε, υποβλήθηκαν από τους σοσιαλιστές ε, και από τη συνάδελφο Μακάρθη 15, 17 και άρθρα 18, 19, 20, 23 και 34 αφορούν μικρές αλλαγές σε σχέση με την προστασία φυσικών ε, προσώπων μετά από τη θέση σε εφαρμογή του πλαισίου αυτού. Η τροπολογία 22 ε, υπερκαλύπτεται από την 1 μετά από ρήτρε διασφάλισης έτσι ώστε να μην υπάρχουν καταχρήσεις ως προς τη διαταγή. Η 34 που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του κανονισμού προτείνει όταν ο λογαριασμός αφορά συγκεκριμένα οικονομικά, χρηματοοικονομικά μέσα, θα πρέπει να ορίζει πού θα ισχύει η διαταγή. Όπως προτείνω και εγώ στην τροπολογία 21, θεωρώ ότι η τράπεζα θα πρέπει να ε, ορίσει σε ποιο χρηματοοικονομικό μέσο ισχύει η διαταγή. Γι' αυτό δεν θα υποστηρίξω αυτή την τροπολογία. Πιστεύω θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε αυτή τη διαδικασία. Θα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες και έτσι νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια πολύ καλή γνωμοδότηση. Θα ψηφιστούν οι προφορικές τροπολογίες στην, στην συνεδρία της ΕΚΟΝ στις 28 Φεβρουαρίου. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε συμβασμό επιθυμείτε. Ευχαριστούμε κύριε Μπασάσκου. Θα ήθελε κάποιος να παρέμβει. Ο κύριος Γκοζές. Τέτοια ώρα. Ένας πρέπει να πει τουλάχιστον ότι ο εισηγητής δούλεψε καλά, τον υποστηρίζουμε και ότι θα ε, ψηφίσουμε με μεγάλη ευχαρίστηση τις τροπολογίες που θα μας προτείνει. Ευχαριστώ και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι η έλλειψη συζήτηση σημαίνει ότι η συγγήτρια έκανε μια θαυμάσια δουλειά και θα έχουμε ευρύτατη και πλατήτατη συνένεση στην ψηφοφορία που θα γίνει στην Επιτροπή ΕΚΟΝ στις 28 Φεβρουαρίου. Τελειώσαμε με αυτά αυτή τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ όλους.